Συναδελφοί, αν θέλετε καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Είναι η πρώτη μας ε, συνεδρίαση με τη νέα χρονιά. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά λοιπόν. Και ελπίζουμε ότι θα είναι για όλους μια καλή χρονιά και για την Επιτροπή μας. Πριν να περάσουμε στην ημερήσια διάταξη, θα ήθελα να σας ε, γνωστοποιήσω ότι έχουμε ένα νέο μέλος ε, στην Επιτροπή που αντικατέστησε την ε, συνάδελφο Γκρούν. Πρόκειται για το συνάδελφο Φιλίπ Μπουρλάν, ο οποίος έχει διοριστεί από το ΕΛΚ. Το καλωσορίζουμε και νομίζω δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Αλλά ήταν ορθό να σας ενημερώσω για την παρουσία του, για την έτου συμμετοχή. Στις περασμένες εβδομάδες έγιναν κάποιες τροποποιήσεις ε, στο σχέδιο ημερησίας διάταξης, το οποίο εγκρίθηκε από τους συντονιστές ε, κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης. Το σημείο 5 που αφορά το follow-up της έκθεσης του Ζωτήλ ε, έχει ανασταλεί για την επόμενη συνεδρίαση γιατί είχε ανελημμένες υποχρεώσεις ο συνάδελφος Μπουζωτήλ το σημείο 7 που αφορά την ανιχνευσιμότητα των αποβλήτων και την ε, σχετικά με το σύστρι έχει ανασταλεί κατόπιν αιτήματος του αναφέροντος. γιατί γίνονται κάποιες συνεννοήσεις με το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην ε, Ιταλία. Έτσι λοιπόν έχουμε αναστείλει την εξέταση. Το σημείο 13 που μια πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών για την έκθεση της Επιτροπής έπρεπε να το αναβάλουμε, αναμένοντας να διοριστεί ο συγητής, ακόμη δεν είχαμε δυνατότητα να το διορίσουμε, αλλά επίσης και ε, λόγω της δημοσίευσης επικαιροποιημένων στοιχείων ε, σχετικά με τις εκθέσεις που παρουσιάστηκαν κατά το 2010, που θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αυτής της ετήσιας έκθεσης. Να σας ενημερώσω ότι προβλέπεται η παρουσία ε, των αναφερόντων ε, στα σημεία 6, 8, 9 και 10 και θα ξεκινήσουμε με αυτή την πρώτη συνεδρίαση. Θα καθορίσουμε τη συνάντηση των συντονιστών όταν θα ολοκληρωθεί ε, η εργασία της Επιτροπής μας. Σήμερα στις 5 θα διακόψουμε τις εργασίες της Επιτροπής μας για να έχουμε τη συνεδρία των συντονιστών και αύριο το πρωί θα ξαναρχίσει η συνεδρία στις 9 με την παρουσία των αναφερόντων για τα σημεία 16, 18, 20 και 21. Πιστεύω αυτές ε, τις ε, αρχικές ανακοινώσεις είχα εγώ από πλευράς μου. Ο συνάδελφος, ε, τον οποίο καλωσορίσαμε την διαποσία του, έφτασε. Εγώ χαιρέτησα συνάδελφε την παρουσία σου και ενημέρωσα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής και κόβεται το μικρόφωνο της Προέδρου για την αντικατάσταση. Καλώς ήρθατε, λοιπόν στην Επιτροπή Αναφορών. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στην έγκριση του σχεδίου της ημερησίας διάταξης. Συνάδελφα, όχι, okay, παρακαλώ. Esauriamo prima questo punto. Eh, Approviamo... Λοιπόν, να εγκρίνουμε πρώτα το σχέδιο τη ημερησίας διάταξη όπω τροποποιήθηκε. Δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Ωραία, θεωρούμε ότι εγκρίνεται λοιπόν το σχέδιο ημερησίας διάταξης. Εγκρίνεται η ημερησία διάταξη. Κύριε Βέρτμαν, για την ημερησία διάταξη, για την έγκριση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση, δηλαδή θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι γίνεται με την ε, ισπανική ε, νομοθεσία για τις ακτές και να το περιλάβουμε στο πρόγραμμα των αναφορών διότι το Δεκέμβριο είχε πει, είχαμε μάθει ότι υπάρχει η νομική αξιολόγηση της νομικής υπηρεσίας οπότε ε, θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται διότι έχω πολλούς Γερμανούς Αυστριακούς αλλά και Ισπανούς υπηκόους οι οποίοι μου στέλνουν επιστολές και μου λέγουν ότι όντως ε, υπάρχει εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας. Ε, πολύ σύντομα ε, θα έπρεπε αυτό όχι μόνο να το περιλάβουμε και να πούμε ότι δεν είναι εξουσιαδοτημένοι για αυτή τη δουλειά αλλά αυτοί όντως συνεχίζουν να πληρώνουν για το ακίνητό τους οπότε ε, έχουν ανησυχίες και θα πρέπει να το συζητήσουμε. Έχουμε όλο και περισσότερους οι οποίοι απευθύνονται σε εμά και θα θέλαμε είτε ε, στην συνέχεια της σημερινής συνεδριάσεως είτε μία από τις προσεχείς συνεδριάσεις να προβλέψουμε και να περιλάβουμε αυτό το θέμα. Ένα λεπτό. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρότασή μου θα ήταν να το συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα στη συνεδρίαση των συντονιστών για να δούμε πώς θα το χειριστούμε και θα δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν. Ωραία, συμφωνώ. Το πρώτο σημείο δεν αφορούσε το έτοιμα τη συναδέλφου. Λοιπόν, κλείσουμε με την έγκριση τη σημερινή ημερησία διάταξη και κατόπιν την παρέμβαση της συναδέλφου θα το δούμε κατά την συνεδρίαση των συντονιστών αργότερα το απόγευμα. Δεύτερο σημείο στην ημερησία διάταξη έγκριση των πρακτικών των προηγούμενων συνεδριάσεων. Όκεν, παρακαλώ. Yes, ε, I... Μάλιστα. Θα ήθελα να πω κάτι για τα πρακτικά της 1ης Δευτέρας Δεκεμβρίου. Να αφηνήσω. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχει κλείσει η αναφορά από τη Ρουμανία. Μπορεί να μην συμφωνείτε, αλλά δεν ε, θεωρώ ότι έχει κλείσει και θα ήθελα να γραφτεί αυτό στα πρακτικά. Και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο εξετάστηκε ήταν ε, μη αποδεκτό από πολλέ απόψει, και θα ήθελα τουλάχιστον αυτό να αναφέρεται στα πρακτικά ότι εγώ δεν θεωρώ ότι έχει κλείσει αυτή η αναφορά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να αναφερθώ στην έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων των ημερομηνιών που αναφέρονται εδώ και αναφέρομαι στα τελευταία πρακτικά ε, να βάλετε και το θέμα του νόμου των ακτών. Εκεί οι συντονιστέ συνιστούν να εξεταστεί αναπερίπτωση το θέμα των αναφορών που έχουμε σε αυτό το νόμο. Εγώ νομίζω ότι δεν συνάδει αυτό με ό,τι υπόθηκε στη συνάντηση των συντονιστών, γιατί όπως θα θυμάστε, πρόεδρος ήσασταν, εκεί υπόθηκε ότι υπήρχε μια πρόταση της κυρίας Βόλης που έλεγε ότι έπρεπε να γίνει αναθεώρηση αναπερίπτωση. Όμως εμείς λέγαμε ότι θα μπορούσαν ε, και άλλες επιτροπές όπως περιβάλλοντος ή νομικών θεμάτων ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιληφθούν. Θα μπορούσαμε εκεί να διαβάσουμε αυτό το θέμα και μάλιστα εμείς ε, ζητούμε και υποστηρίζουμε την παρουσία του Ισπανού διαμεσολαβητή, του συνηγόρου του πολίτη. γιατί καθώς εδώ έχουμε θέματα ε, τα οποία συστήνουν οι συντονιστές αναπερίπτωση να εξεταστεί αυτός ο νόμος. Εγώ επαναλαμβάνω ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και θα το δούμε αυτό και στη συνέχεια στη συνεδρίες των συντονιστών. Έτσι λοιπόν, καλό είναι να σημειωθεί εδώ το τι υπόθηκε στη συνεδρίαση των συντονιστών τότε και όχι η πρόταση της κυρίας Γκόλης ε, να παρουσιάζεται ως πρόταση όλων των συντονιστών. Κολέγα Μποστινάρου. Μποστινάρου. În condițiile în care au fost discuții între coordonatorii grupului. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, δεδομένου ότι υπάρχει συζήτηση μεταξύ των ε, συντονιστών των ε, πολιτικών ομάδων για την αναφορά που αφορά την ε, ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στη Ρουμανία και δεδομένου των συμβιβασμών στους οποίους καταλήξαμε μετά από τις διαπραγματεύσεις, σας προτείνω στα πρακτικά της τελευταίας μας συνεδρίασης να γίνει μια αναφορά στην ε, ε, συγκεκριμένη αναφορά από την Ρουμανία. Σήμερα στους συντονιστές θα επανέλθουμε ή δυνατόν στη συγκεκριμένη αναφορά και νομίζω ειλικρινά ότι πρέπει να καταλήξουμε σε μία λύση που να μπορεί να εξασφαλίσει τα συμφέροντα και της δικής μας ε, Επιτροπής. είτε αύριο πρέπει να το συμπεριλάβουμε στην ημερήσια διάταξή μας, είτε στην επόμενη συνεδρίαση. Και το λέω αυτό συμβιβαστικά για να μπορέσουμε να εξετάσουμε και αυτή την αναφορά και να ε, μπορέσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, εγώ ήθελα να αναφερθώ σε κάτι σχετικά με τα διάφορα. Μάλιστα, δεν έχει ζητήσει κανεί άλλο το λόγο. Επομένω, πιστεύω ότι για το θέμα τη έκθεση των πρακτικών των προηγούμενων συνεδριάσεων μπορώ να προτείνω να εγκρίνουμε τα πρακτικά τη 9η Νοεμβρίου και τη 22η Νοεμβρίου, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Και για τη συνεδρίαση 1η και 2η Δεκεμβρίου. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι έκαναν κάποιες παρατηρήσεις που πήραν το λόγο και οι τρεις συνάδελφοι. Προτείνω λοιπόν να ψηφίσουμε την έγκριση των πρακτικών αύριο το πρωί. Αφού θα έχουμε συζητήσει σήμερα το θέμα αυτό στη συνεδρίαση των συντονιστών. Να συγκρίνουμε λοιπόν τα δύο πρώτα πρακτικά και αύριο το πρωί θα ψηφίσουμε για τη συνεδρίαση 1η 4 Δεκεμβρίου. Σε ό,τι αφορά τώρα το σημείο 3, ανακοινώσει. Πρέπει να σα κάνω κάποια ανακοινώση σε σχέση με τι σημειώσει που υπάρχουν για το δεύτερο τμήμα τη ημέρης τη διάταξη, ε, όπου έχουν εγγραφεί αναφορέ ε, ε, που προτείνονται για να εξεταστούν και για να κλείσουν, ανάλογα με τι προτάσει των διαφορών συναδέλφων. Έτσι λοιπόν, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ε, για το τμήμα αυτό, εγκρίνεται έτσι όπως βλέπετε τα στοιχεία στην πρόταση που έχει διανεμηθεί στους συναδέλφους. Λοιπόν, στα διάφορα, συναδέλφους Μπίλαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να υποφεληθώ της ευκαιρίας να προτείνω κάτι το οποίο έχω ε, απευθύνει επανειλημμένος γραπτό στη γραμματεία. Δηλαδή έχουμε ε, συνοπτικές παρουσιάσεις από πολλαπλές αναφορές και η πρότασή μου αναφέρεται στην περαιτέρω διαδικασία διότι συνήθως δεν έχουμε αρκετό καιρό. Ε, τα χρονικά περιθώρια είναι περιορισμένα, δεν έχουμε αρκετό χρόνο να υποβάλουμε γραπτός ε, προτάσεις και ήθελα ήθελα να σας πω και με ενδιαφέρει πολύ αυτό εις ε, την ε, προθεσμία να περιλαμβάνει κανείς μέχρι την επόμενη συνεδρίαση ώστε αν δεν υπάρχει ένα γραπτό, μια γραπτή αιτιολογία να μπορεί να αναφερθεί οτιδήποτε ή στα πρακτικά και αυτό είναι πολύ ουσιαστικό για τις διαδικασίες. Ε, θα ήθελα να παρακαλέσω. Αν ε, παραδείγματο χάρη να έχουμε τη μετάφραση στις 15 του μηνός ή χρειάζονται 10 μέρες και μετά η πρώτη συνεδρίαση είναι στην πρώτη του μηνός και εάν είναι πολύ κοντά η δεύτερη τότε μπορούμε να περιμένουμε μέχρι την τρίτη. Δηλαδή να βάλουμε πιο μακριές προθεσμίες για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί δεν είναι καλό το παρόν σύστημα, δηλαδή απευθύνουμε ε, γραπτός ηλεκτρονικά μηνύματα στην ε, γραμματεία και μετά κύριε ε, θα ήθελα να, να μου απαντήσουν τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να προχωρήσει το θέμα. Ενώ έτσι όπως πάμε τώρα δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό το σύστημα. Συνάδελφε, αν κατάλαβα καλά, η πρότασή σας είναι να μην θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα της ημερησίας διάταξης, το τμήμα Β δηλαδή, τότε δεν σας κατάλαβα. Τα έγγραφα διανεμήθησαν. Πάντοτε έχουμε 20-25 αναφορές και έχουμε ε, συνοπτικά την παρουσίαση, τις, τα συμπεράσματα και ε, τις αποφάσεις. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία ε, διεκπεραιώνονται και ετοιμάζονται πριν από την ημερομηνία της Επιτροπής. Συνήθως ο βουλευτής έχει 4, 5, 6 μέρες και πολλές φορές ακόμη λιγότερο ή καθόλου και ήθελα να σας πω ότι εμένα δεν με ικανοποιεί αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, προτού τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή πριν από τρεις, τρεις μήνες πριν από το δεύτερο τμήμα, νομίζω ότι θα είχαμε καιρό να ασχοληθούμε με αυτό το χαρτί και θα ήθελα να έχουμε μια καλύτερη διαδικασία. Δεν μου ήταν σαφές. Γιατί εσείς υπογραμμίζετε το ότι μας πίζει ο χρόνος, ότι δεν υπάρχει της προθεσμία μεταξύ της ε, αποστολής αυτού του εγγράφου, που αποκαλείται ΣΥΡ, και της ε, δυνατότητας να προγραμματίσουμε ε, τις αιτήσει αυτές, τις αναφορές αυτές. Υπάρχει ένα πρόβλημα λοιπόν. Τα έγγραφα στέλνονται στους συναδέλφους αφού έχουμε λάβει έναν αριθμό αναφορών και που να έχουν εξεταστεί από την γραμματεία και που να φέρουν και μία γνωμοδότηση επί της ουσίας κάθε μέλος μπορεί να εκφράσει τη δική του θέση. μέσα σε κάποιες μέρες από τη στιγμή που έχει ληφθεί το σύνολο αυτών των αναφορών. Στη συνέχεια ε, τι τίθεται σε πρόγραμμα εξέτασης ανάλογα με την αξιολόγηση που θα έχει γίνει. Έτσι λοιπόν εσείς ζητάτε να μην επιμικίνουμε αυτή την προθεσμία από την αποστολή μέχρι τον προχρηματισμό που είναι κάτι που ενδεχομένω θα γίνει στο μέλλον. Θέλετε να έχουμε περισσότερο χρόνο, το χρόνο που δίνεται στο κάθε μέλος για να κάνει τη δική του αξιολόγηση επί της πρότασης που έχει διατυπωθεί. Δηλαδή αντί για τρεις μέρες να έχουμε πέντε μέρες. Δηλαδή να επικίνουμε το χρόνο για την αξιολόγηση. Νομίζω ότι και αυτή είναι μια πρόταση που μπορούμε να τη συζητήσουμε με τους συντονιστές. Ας το θέσουμε και από τα διάφορα και για σήμερα, αν μπορέσουμε να εξαγγελίσουμε και αυτό το θέμα. Θα προσπαθήσουμε να λάβουμε υπόψη το αίτημα να υπάρχει μεγαλύτερη προθεσμία για να μπορούν να εξετάζονται όλες οι προθέσεις που διατυπώνονται με τα έγγραφα αυτά. Πολύ. Εντάξει, groben. Σε γενικές γραμμές, ναι, κυρία Πρόεδρε. Αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν καταλαβαίνω αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, στην αρχή ε, η γραμματεία ε, έχει μία συμπεριφορά ε, όπου δεν εμπλέκεστε και εάν η γραμματεία συμφωνεί με την πρότασή μου πρέπει η γραμματεία να συζητήσει το θέμα μαζί σας και αυτό δεν έχει γίνει. Δεν αναφέρομαι στα 8 ηλεκτρονικά ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία έχω απευθύνει στη γραμματεία μέχρι στιγμής, αλλά θα τους παρακαλούσα να σας ενημερώσουν περί τίνος πρόκειται. Για το δεύτερο τμήμα της παρέμβασής σας. Σίγουρα θέτει ένα ερώτημα το οποίο αναλαμβάνω εγώ. Ευχαριστώ να λάβω από σας ε, όλα τα έγγραφα σε αντίτυπο τα έγγραφα που αποστέλλονται στην, στην Επιτροπή. Συμφωνώ απόλυτα, γιατί είναι προφανές ότι οι γνωμοδοτήσεις ε, των βουλευτών για τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη δεόντως, γιατί διαφορετικά ματαιώνεται η διαδικασία. Αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να ενημερωθεί η Προεδρία έτσι ώστε να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να αποφευθεί οι αξιολογήσεις και θέσεις των συναδέλφων να έχουν αξιολογηθεί δε Τώρα, αν ε, εσείς ε, μου πείτε ποιοι είναι οι συνάδελφοι που θέλουν να λαμβάνουν τις απαντήσεις σε αντίγραφο, τότε δεν υπάρχει καμία αντίρρηση για τη συνεδρίαση των συνεστών να προσπαθήσουμε να αστήσουμε πιο αποτελεσματική τη διαδικασία. Ας περάσουμε στο επόμενο σημείο και ας ξεκινήσουμε με την εξέταση των αναφορών. Ας περάσουμε απευθεία στο σημείο 6 της κυρία Μαρία Γκράτσα Κανούτη για το χώρο διάθεση αποβλήτων στη Μαλαγκρότα κοντά στη Ρώμη. Η κυρία Κανούτη θα πρέπει να είναι παρούσα. Κυρία Κανούτη, καταρχήν έχει το λόγο. Pronto? Ok. Um, allora, io... Εγώ σας έχω φέρει για κάποιες φωτογραφίες για να εξηγήσω καλύτερα την κατάσταση. Το 1955 ο πατέρας μου πήγε να δουλέψει στη Ρώμη και σε κάποια λεωμέτρα που βρισκόταν 18 χιλιόμετρα από την ακτή της Τουρνίας και 13 χιλιόμετρα από το Καπιτόλιο. Εδώ μπορείτε να δείτε τις αποστάσεις. Το 1978 ε, κατασκευάσαμε ένα νέο σπίτι, 55 μέτρα σχεδόν από ε, αυτή την τοποθεσία των σπιτιών σε μια νέα ε, ζώνη ανάπτυξης, κατασκευαστικής ανάπτυξης, η οποία αναπτυσσόταν βάσει συμφωνιών με το Δήμο της Ρώμης. Εμείς ε, μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση σε πηγάδια για το πόσιμο νερό και ε, ε, μπορώ να σας πω ότι είχαμε καθαρό αέρα και πολύ καλές θερμοκρασίες γιατί βρισκόμασταν αρκετά κοντά στη θάλασσα η οικογένεια μου ε, από το 78 και μετά ε, αναγκάστηκε να πληρώνει τις επιχειρήσεις, την κοινοπρεξία για τις επιχειρήσεις, μάλλον τις υπηρεσίες όπως ήταν ε, το πόσιμο νερό, η διατήρηση των δρόμων, γιατί δεν προσφέρονταν ακόμη από το Δήμο, αλλά και το Δήμο της Ρώμης για κάποιους φόρους. Έπρεπε να χορηγηθούν χρήματα για κάποιους φόρους. Με συγχωρείτε, έκανα λάθος λέει μιλήτρια. Τότε, το 1978, σε μια περιοχή που δεν ήταν δυνατό να μετατραπεί σαν κρατομαχία, ένας ιδιοκτήτης, ο ιδιοκτήτης μάλλον, ε, της τοποθεσίας αυτής, άρχισε να χρησιμοποιεί το έδαφος αυτό ως ε, παράνομη χωματερή. Και υπήρχαν ε, ε, διαμαρτυρίες ε, γιατί ήδη το 78 ήταν ιδιαίτερα κατοικημένη αυτή η περιοχή ε, Επρόκειτο για τις περιοχές Μαλαγκρότα και Μασιμίνα. Εκεί είχαμε περιοχές όπου είχαμε ε, και αρχαιολογικά ευρήματα και ε, σε αυτό το κίτρινο σημείο, τετράγωνο, βλέπετε με κόκκινο που βρισκόταν ε, το σπίτι μου. Και εμείς ήμασταν 1,5 χιλιόμετρο από από αυτή την παράνομη χωματερή. Το 1984 η κοινότητα, ο Δήμος της Ρώμης, ε, καταρχήν ε, καταναγκαστικά, ε, μάλλον εξαιρετικά, αλλά στη συνέχεια πιο συχνά άρχισε να χρησιμοποιεί αυτή τη χωματερή για τα αστικά απόβλητα άρχισε μάλιστα να τη χρησιμοποιεί κάποτε και καθημερινά. Το 1990 ο πληθυσμός της περιοργής άρχισε να διαμαρτύρεται. Εδώ βλέπετε δύο μαύρες κουκίδες, ε, βλέπετε ε, πώς έχει επεκταθεί η χωματερή Βλέπετε εδώ αυτό το κομμάτι που ξεκινά από την Οδό Ουρέλια όπου λέει Κασάλου Λουμπρόζο. Έχουμε περίπου 3,5 χιλιόμετρα. Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε πόσο μεγάλη είναι αυτή η χωματερή, αυτός ο χώρος διαθέσεις αποβλήτων. Εγώ δεν ε, μπορώ να την μετρήσω με τεχνικά μέσα, αλλά είναι πολύ μεγάλη. Ο μόνος δήμαρχος ε, που έκανε κάτι είναι να υπάρχει ένας χώρος πρασίνου, μάλλον δύο χώροι πρασίνου μπροστά στην ε, χωματερή βλέπετε με μοβ ε, περιοχές ε, εκεί έχουν δημιουργηθεί κάποιοι χώροι δίσοσμοι. Εγώ υποθέτω ότι ε, είναι λόγω της το συγκοινωνούνταν δοχείων, δηλαδή κάποια απόβλητα κάποια λίματα φεύγουν από τη χωματερή και καταλήγουν σε αυτούς τους τόπους. Ε, βλέπετε στη συνέχεια ε, το 2010 άνοιξε μια χαράδρα στην πρώτη κουκίδα και το 2009 υπήρξε μια κατολίσθηση. Δηλαδή εκεί ε, έφυγαν τα σκουπίδια και έπεσαν στο δρόμο και έγινε μια παράκαμψη της κυκλοφορίας εκεί και ο αρχικός δρόμος δεν υπάρχει πια. Λοιπόν, ε, πώς ε, κατασκευαστήκε αυτό το τέρας. Ε, καθημερινά φτάνουν φορτηγά που τοποθετούνται στις άκρες αυτού του βουνού μπροστά σε μπουλντόζες και ε, συνδέονται με ρημουλκά και ε, σέρνουν αυτά τα, τα απόβλητα και στη συνέχεια αναλαμβάνουν τη δουλειά οι μπουλντόζες. Και πάντοτε έχουμε σωματίδια στην περιοχή, έχουμε δυσοσμία και αυτές οι ουσίες ε, διαδίδονται και με τον άνεμο. Και φυσικά φαντάζεστε τι, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει όταν έχουμε υψηλέ θερμοκρασίε. Εγώ αρρώστησα το 2006 αφού είχαμε καλοκαίρι με υψηλέο ε, με υψηλές θερμοκρασίες ε, βλέπετε ότι αρρώστησα και στη συνέχεια είχαμε τα στάσεις στο στομάχι στο σηκώτη και στα γενετικά όργανα. Ε, αυτό που βλέπετε έχει δημιουργηθεί από μία συσσόρευση υγρών από τα αντισώματα των οργάνων στα οποία επιτίθεται η μετάσταση του καρκίνου. Ε, εγώ υπέστησα τη χημειοθεραπεία από το Σεπτέμβριο του 2008 μέχρι το Φεβρουάριο του 2009 με έξι επαναλήψεις που διέρχεσαν η κάθε μία οκτώ ώρες. Ο γιατρός ε, δεν ε, θεώρησε ότι έπρεπε να με θεραπεύσει και από τη συνέπειες της χημειοθεραπείας. η χημειοθεραπεία σταμάτησε την αναπαραγωγή των καρκινογόνων κυτάρων, αλλά αποδυναμώθηκε το, το σύστημα, τον, ο σκελετός μου, μου πέφτουν τα δόντια, πάσχω από ισχυρή οστεοπόρωση, έχω προβλήματα ε, με την όρασή μου και χάνω την ισορροπία μου. βλέπετε ότι αυτό το πρίξιμο ε, πιέζει τα υπόλοιπα όργανα, το στομάχι, την καρδιά, τα έτερα, ε, του, τα, νεφρά, τους ε, πνεύμονες. Αυτό προκαλεί σε μένα δυσκολίες να κοιμηθώ, έχω ναυτίες, μετούς, κουράζομαι πάρα πολύ, και είναι αδύνατο για μένα να έχω μια φυσιολογική ζωή. Έτσι λοιπόν εγώ θεωρώ υπεύθυνος για το έγκλημα αυτό ε, όσους θα έπρεπε να ελέγχουν ε, το περιβάλλον σε αυτή την ε, περιοχή. Θεωρώ όσους διακυβέρνησαν τη Ρώμη από το 67 ως ε, το 76 γιατί δεν σχεδίασαν και δεν ξεκίνησαν εργασίες για την ορθή διάθεση των αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους. Και ε, οι δήμαρχοι που ήταν... που, κυβερνούσαν την πόλη από το 1976 στο 2011 είναι επίσης υπεύθυνοι γιατί ε, έχουν ε, εμπιστευτεί μία τόσο επικίνδυνη ε, χώματερη όπου έχουμε κάθε είδους απόβλητα, νοσοκομιακά, βιομηχανικά απόβλητα σε κάποιον που είναι ανίκανος να τα διαχειρίζεται και μάλιστα έχουν επιτρέψει να υπάρχει αυτή η χωματερή μόνο 13 χιλιόμετρα από το Καπιτόλιο, σε μια ζώνη ιδιαίτερα κατοικημένη. Με συγχωρείτε, ολοκληρώθηκε ο χρόνος μου. Λοιπόν, επίση άλλη υπεύθυνη είναι όσο από το 1978 στο 2011 ε, δεν διαχειρίστηκαν ε, σωστά τις ε, ποσοστώσεις σε σχέση με τη γη. Και επίσης υπεύθυνο είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου της χωματερής, ο οποίος έχει εμποδίσει κάθε έργο ανάκτησης και ανακύκλωσης ε, των αποβλήτων με αποτέλεσμα να έχουμε παραγωγή αερίων σε βιομηχανικό επίπεδο. Και εγώ αναρωτιέμαι γιατί αγνοώ πόσα υλικά και μάλιστα δοξικά χρησιμοποιούνται ε, για να μετατραπούν ε, σε αέρια τα απόβλητα, πόσες τοξικές ουσίες παράγονται από ένα λίτρο αερίου από τα απόβλητα και πού αυτά τα απόβλητα θα ε, αποθηκευτούν, θα πρέπει να παραμείνουν ε, μπροστά στο σπίτι μου για πολύ καιρό ακόμη. Πρέπει να ολοκληρώσετε. Ήθελα απλά να σας δείξω κατακόμη Αυτό το 2006 βλέπετε ότι αυτό το τέρας ε, ξεπέρασε τη γραμμή του ορίζοντα. Εδώ βλέπετε τους λόφους γύρω-γύρω και εκεί βλέπετε τη χωματερή. Εδώ το 2010 ε, βλέπετε μέχρι που φτάνει και το 2011 βλέπετε πόσο έχει μεγαλώσει σε σχέση με το 2010. Εγώ δεν βλέπω πια τον ορίζοντα, βλέπω μόνο αυτό το βουνό από σκουπίδια. Τελείωσα και σας ευχαριστώ. Grazie. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Έχει ήδη ξεκινήσει με έρευνα για την καταγγελία ε, της αναφέρουσας. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Γιώργο Κουδέσκου. Thank you, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως είπατε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει η έρευνα για τη διαχείριση της ε, χωματερής της ε, Μαλαγκρότα μετά από ανταλλαγή απόψεων ε, με τις Ιταλικές αρχές. Ζητήθηκε μία Έγινε μια νέα αίτηση για περαιτέρω πληροφορίε τον Ιούνιο του 2010. Από τότε το θέμα ήταν αντικείμενο πολλών επαφών μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ιταλικών Αρχών και μάλιστα σε σχέση και με μία άλλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά το νέο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για την περιοχή του Λάτσιο η έγκριση του οποίου αναμένεται στο πρώτο ήμιση του 2011. Η έρευνα για το πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων του Λάτσιο είναι βέβαια διαφορετικό θέμα, ξεχωριστό φάκελο και έχει ξεκινήσει ήδη μια διαδικασία επίσημη επί παραβάση, ενώ το θέμα της Μαλαγκρότα είναι μια προκαταρκτική έρευνα. Η σχέση μεταξύ των δύο θεμάτων είναι ότι το πρόγραμμα του Λάτσιο πρέπει να αφορά όλους τις χωματερές και τις Μαλαγκρότα. Σε πρόσφατη συνεδρίαση την περασμένη εβδομάδα για το νέο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων του Λάτσιο, ε, που είχαν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις Ιταλικές Αρχές, υπενθύμησε η Επιτροπή στι Ιταλικέ Αρχέ ότι πρέπει να αποστείλουν μια επίσημη απάντηση σε αυτή τη νέα αίτηση περαιτέρω πληροφοριών ε, για ε, το θέμα της Μαλαγκρότα. Η απάντηση των Ιταλικών αρχών ε, στα ερωτήματα που αφορούν τα ζητήματα στα οποία αναφέρεται η κυρία Κανούτη αναμένονται σύντομα από τις Ιταλικές Αρχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει τα στοιχεία αυτά για να δει κατά πόσο υπάρχει μια παραβίαση του ισχύοντος περιβαλλοντικού νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως το είπα, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ένα ευρύτερο θέμα, είναι τμήμα ευρύτερου θέματος ε, του προγράμματος ε, διαχείρισης αποβλήτων ε, του Λάτσιου που αφορά βέβαια και την διαχείριση της κομματερής της Μαλαγκρότα. Ευχαριστώ. Αναμένουμε λοιπόν ακόμα την απάντηση των ε, τοπικών αρχών. Ε, η Επιτροπή πάντως έχει αναλάβει δράσεις ε, επί του θέματος. Συνάδελφος ο Τουρκάη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αφού άκουσα τα όσα μας είπε η αναφέρουσα, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι είναι ανατριχιαστικά τα όσα ακούσαμε γιατί εδώ μιλάμε για ανθρωπίνες ζωές. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι απέναντι σε αυτή την αναφορά. Και αφού ακούσαμε για την Επιτροπή, είναι σαφές ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε, πρόεδρε, είναι να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά, γιατί αν εδώ και επτά μήνε που έχουμε ζητήσει τις ε, πληροφορίες δεν έφτασαν ακόμα και η Επιτροπή, η Κομισιόν ε, παραπονιέται, γιατί δεν έχουν σταλεί ακόμα τι πληροφορίε, ε, θα μα πει η Κομισιόν ότι τελικά χρειάζεται αυτέ τι πληροφορίε για να μπορεί να καταλήξει κάποια απόφαση. Έτσι λοιπόν μέχρι να έλθουν οι πληροφορίε, εγώ θα αφήνα ανοιχτή την αναφορά και ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή τις επόμενες ώρες ε, και όχι μέρες να έλθει σε επαφή με τις Ιταλικές αρχές για να ζητήσει αυτές τις πληροφορίες. Γιατί επιμένω, ήδη έχει περάσει πάρα πολύ καιρό, μιλάμε για 7 μήνες. Δηλαδή μια πληροφορία ζητήθηκε, αλλά μπορεί να μας διευκρινίσει η Κομισιόν. Μία φορά ζητήθηκαν οι πληροφορίες ή πολλές φορές επιμείνατε να σας στέλνω σε αυτές τις πληροφορίες, γιατί μέσα σε 7 μήνες πολλές φορές ε, θα μπορούσατε να τις είχατε ζητήσει για να τις έχετε σήμερα. Τώρα είδαμε 7 μήνες μετά ότι έπρεπε να έρθει η αναφέρουσα στη δική μας επιτροπή εδώ στις Βρυξέλλες. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ενδεχομένως να μην άκουσα πολύ καλά. Αλλά δεν πρόκειται για τις περιβαλλοντικές οδηγίες, πρόκειται επίσης και για τις οδηγίες περί αποβλήτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και θα ήθελα να μάθω κατά πόσο προτιθέμεθα να λάβουμε υπόψη το ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η οδηγία για τα απόβλητα. Μου έκανε όμω εντύπωση γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν αναφέρθηκε. Μιλήσαμε μόνο για τι οδηγίε για το περιβάλλον και όχι για τι οδηγίε για τα απόβλητα. Θα ήθελα λοιπόν να είμαι απολύτω βέβαιη ότι θα ληφθεί υπόψη και η οδηγία περί αποβλήτων. Ευχαριστώ. Υπάρχουν τρία θέματα. Είναι οι οδηγίες για τα σκουπίδια και ε, συγκεκριμένα ιδίω για την υγεία των ανθρώπων. Οπότε με ενοχλεί πάρα πολύ που η διαδικασία αυτή κρατά τόσο καιρό. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να πούμε ότι και να έρθει αργότερα η πληροφόρηση δεν μας πειράζει. Νομίζω ότι εδώ υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις και ο ετών έχει το δικαίωμα να έχει μία σύντομη απάντηση. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόσο γρήγορα αναμένει ότι θα έχει μία ικανοποιητική απάντηση από τις ε, Ιταλικές ε, ε, αρχές. Μέχρι τότε θα αφήσουμε ανοιχτό το θέμα αλλά δεν βοηθάμε εδώ την ετούσα η οποία θα ήθελε μία ικανοποιητική απάντηση είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε από τις Ιταλικές Αρχές. Παρακαλώ, έχετε το λόγο μου πώς μπορείτε να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Όπως είπα και προηγουμένως, είναι θέμα επίγον και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τις υπηρεσίες της. Ε, γνωρίζουμε ότι έχουν περάσει 7 μήνες από τότε που κάναμε την τελευταία αίτηση για περαιτέρω πληροφορίες και όπως είπα είχαμε και διμερείς επαφές από τότε με τις Ιταλικές αρχές. Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα και συμφωνώ με τους συναδέλφους σας ότι καλύπτει μεγάλο τμήμα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της απόθεσης αποβλήτων. Κάτι το οποίο βέβαια η κακή εφαρμογή δηλαδή έχει, κάτι, έχει επιβλαβεί συνέπειες ε, στην ανθρώπινη υγεία. Όπως είπα την περασμένη εβδομάδα, την Πέμπτη συζητήσαμε με τις Ιταλικές Αρχές και περιμένουμε την απάντησή τους πολύ σύντομα. Και μόλις λάβουμε την απάντηση αυτή θα κάνουμε και τα επιπλέον ε, βήματα. Ελπίζουμε ότι θα είναι ικανοποιητική η απάντηση των Ιταλικών αρχών ή αν δεν τη λάβουμε, έχουμε κάποια νομικά μέσα στη διάθεσή μας και όπως είπα ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει το θέμα αυτό ως κατεπήγον. Και όπως είπα, επίσης, σε σχέση με το πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων του Λάτσιο, είναι και το θέμα της απόθεσης των αποβλήτων. Δεν αφορά μόνο το θέμα της ε, Μαλαγκρότα, δεν επηρεάζεται μόνο η Μαλαγκρότα δηλαδή, αφορά ολόκληρη την περιοχή ε, Λάτσιο. Οπότε συνεργαζόμαστε με τις Ιταλικές Αρχές και ελπίζουμε κατά τις ερχόμενες εβδομάδες ε, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Eh, Σας ευχαριστώ. Πιστεύω ότι από την πλευρά όλων υπάρχει συμφωνία ότι πρέπει να συνεχίσουμε και να προωθήσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό, γιατί δεν λάβαμε απάντηση από την Επιτροπή, γιατί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει λάβει απάντηση από τις Ιταλικές Αρχές. Έτσι λοιπόν είναι επίγουσα η κατάσταση και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρέπει να επευθυνθούμε και πάλι στις Ιταλικές αρχές. Ίσως θα μπορούσαμε και εμείς να, να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία, να επευθυνθούμε στις Ιταλικές αρχές. Δηλαδή και εμείς θα μπορούσαμε να καλέσουμε τις Ιταλικές αρχές σε μία κρόση ή να ζητήσουμε μία επίγουσα απάντηση. Και αν ε, είχαμε και μία θετική απάντηση για την παρουσία των τελικών αρχών εδώ στην Επιτροπή μας, ε, θα μπορούσαμε την επόμενη φορά να το προγραμματίσουμε έτσι ώστε για να ακούσουμε τις Ιταλικές αρχές αν αποφασίσουν να παραβρεθούν. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια δυνατότητα. Και κατόπιν θέλω να ζητήσω, να ρωτήσω την αναφέρουσα αν θέλει κάτι να προσθέσει. Έχετε κάποιο σχόλιο επιπρόσθετο. Έχετε λίγα λεπτά. Κοιτάξτε, η τελευταία είδηση ήταν ε, ότι ε, ο Δήμαρχος και ε, ο Νομάρχης έριχναν τον μπαλάκι ο ένας στον άλλο να βρουν ο μία λύση. Το πρόβλημα μου όμως είναι τι θα κάνω εγώ με αυτό το τεράστιο βουνό από σκουπίδια μπροστά από το σπίτι μου γιατί συνεχίζουμε να αναπνέουμε αυτή τη σκόνη και φοβάμαι ότι, ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται ο όγκο των σκουπιδιών και να μεγαλώνει όλο ένα και περισσότερο το βουνό και με αυτές τις εγκαταστάσεις που θέλουν να φτιάξουν για την ε, επεξεργασία. Πρόεδρος, ε, κοιτάξτε, εμείς ε, δεν μπορούμε να σας δώσουμε μια απάντηση αυτή τη στιγμή. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε άμεσα είναι να σας βοηθήσουμε να σας δοθεί απάντηση από τις αρμόδιες αρχές, δηλαδή από το Δήμαρχο και από το Ονομάρχη από τον Περιφερειάρχη. Εμείς ε, ζητήσαμε όχι μόνο από την Εκτελεστική Επιτροπή να ζητήσει μια μέση απάντηση από στα αιτήματα που έχουν διατυπωθεί, αλλά και εμεί θα δραστηριοποιηθούμε ω Επιτροπή Αναφορών για να ζητήσουμε από τον Περιφερειάρχη και από τον Δήμαρχο να έλθουν εδώ οι αντιπροσωποί του και να μα δώσουν κάποιε απαντήσει και να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς ε, σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που υπάρχει και πότε γιατί δεν θα ήθελα και να υπάρχει ένα άλλο τεράστιο τέρας κάπου αλλού μια άλλη παρόμοια χωματερή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Παστινάρη. Ε, uh, Θα ήθελα να υποστηρίξω την πρότασή σας κυρία Πρόεδρε. Για δύο λόγους. Πρώτον, είναι προφανές ότι εμείς ως Επιτροπή Αναφορών πρέπει να κάνουμε κάτι για την αναφέρουσα. Δεύτερον, Νομίζω ότι έχουμε δει τόσες πολλές, φορές, τόσες πολλές τέτοιες υποθέσεις ε, επανειλημμένως που οι εθνικές κυβερνήσεις είτε αρνούνται να απαντήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή καθυστερούν τόσο πολύ, περνάνε χρόνια και χρόνια μέχρι να απαντήσουν ενδεχομένως να γίνει μια ειδική συνάντηση με τον Επίτροπο Σεύτσοβιτς που είναι ο υπεύθυνος για, το, ε, για, τις, ε, για την διαθεσμική συνεργασία για να δούμε πώς μπορούμε να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα, χρονοδιάγραμμα στις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ξέρω τι είδου συντονισμός ε, θα χρειαστεί, τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε, αλλά Είναι πραγματικά ντροπή οι κυβερνήσεις να μην απαντούν. Γιατί πραγματικά αυτό συνιστά έλλειψη συμβασμού, ε, σεβασμού και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το να σημειώνουμε απλώς αυτή την ε, συμπεριφορά είναι τελείως απαράδεκτο. Σας ενθαρρύνω πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, να στείλετε αυτή την επιστολή στην Ιταλική κυβέρνηση, όπως επίσης και να γίνει και η συνάντηση με τον Επίτροπο Σεύτσοβιτ, τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να βρούμε έναν τρόπο. Μία λύση βιώσιμη, γιατί διαφορετικά είμαστε άχρηστοι. Σε πολύ συγκεκριμένε περιπτώσει είμαστε πάρα πολύ, είμαστε άχρηστοι στο να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την υγεία και τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Συνάδελφο Γιάρσε. Ε, θέλω να στηρίξω το θέμα διότι αυτό είναι το ουσιαστικό πρόβλημα για την Επιτροπή Αναφορών. Αν δεν έχουμε ενημέρωση για τα κράτα, από τα κράτη-μέλη δεν μπορούμε να αποφανθούμε για την αναφορά. Δεν αναφέρουμε εδώ στη συγκεκριμένη αλλά έχουμε πάρα πολλές αναφορές που αναφέρονται στα θέματα περιβάλλοντες και πολλές ε, φορές ε, εσχεμένως οι κυβερνήσεις καθισταυρούν ότι ε, εάν αργήσουμε και καθυστερήσουμε δεν θα μπορεί να αλλάξει τίποτα ως προς τα ουσιαστικά στοιχεία. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια συμφορία κυρίων ή κάποιο σύστημα σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να λαμβάνουμε απαντήσεις γιατί βλέπω σε πάρα πολλές αναφορές την τελευταία φράση να αναφέρεται ότι οι τελευταίες απαντήσεις από το κράτος μέλος απλώς απουσιάζουν. Κάποια στιγμή έτσι δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική γνώμη του θέματος. Ευχαριστώ. Παραμένει ανοιχτή λοιπόν η αναφορά στο στάδιο αυτό. Η Προεδρία αναλαμβάνει να απευθυνθεί στις αναλογοαρχές για να τις προσκαλέσει να πρευρεθούν εδώ στην Επιτροπή ή να στείλουν μια επίγουσα απάντηση. Και Φυσικά, καλό και την Κομισιόν να επιταχύνει τις διαδικασίες για την απόκτηση των απαντήσεων στις ερωτήσεις που έχουν τεθεί. Ευχαριστώ την αναφέρουσα και θα περάσω στο επόμενο σημείο την αναφορά που παρουσιάστηκε από τον κύριο Κράστε, Φιβέλο Συνοφ θα πρέπει να είναι παρόν. Θα ήθελα να του δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να σας συστηθώ. Λέγομαι Βέσισλαφ Μπουζίλουφ, είμαι ο πρόεδρος ε, του κινήματος προστασίας ε, της υγείας ε, των κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής. Πρόκειται για την αναφορά 1405 του 2007 σε σχέση με τα προβλήματα της συνοικίας Σουοντόλ στη Σόφια. Κυρία Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, ε, θα σας παρουσιάσω την άποψη των κατοίκων της περιοχής μας και ειδικότερα σε σχέση με την εκμετάλλευση μιας παράνομης χωματερής ε, της ε, περιοχής Σουχοντόλ. Κατόπιν ετήσεως της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υποβάλαμε έγγραφα, όπως επίσης ε, και βίντεο, σε σχέση με την ε, οδηγία 12 του 2006 ε, και η 98 του 2008 δεν έτυχαν, δεν, έγι, δεν έτυχαν σεβασμού. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό γιατί γίνεται παραβίαση της, ε, της οδηγίας 2060 ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, για τα ύδατα, δεδομένου ότι σε υπόγεια ύδατα ε, καταλήγουν τελικά τα απόβλητα που εναποτίθενται. Πρόκειται λοιπόν για μεγά, πολύ σοβαρές παραβιάσεις και πολύ ε, κακές συνέπειες για την υγεία των ε, κατοίκων. Πολλές φορές ε, ζητήσαμε να γίνει μια επίπτωση, μια εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όμως δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο. Υποθέτω ότι έχετε ήδη υπόψη σας τα, το υλικό που υπήρξε από βίντεο και παρουσιάστηκε και στην τηλεόραση. Προς την, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, απευθύνθηκε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών ε, Κοινοτήτων και ε, κατηγόρησε τη Βουλγαρία ότι δεν έχει προβλέψει κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων, για την επεξεργασία τους. Ε, ήταν πολύ σαφές λοιπόν ότι οι βουλγαρικές αρχές εξακολουθούν ε, να χρησιμοποιούν, εκμεταλλεύονται την παλαιότερη χωματερή του Σιχοντόλ, του Σιχοντόλ που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται μάλλον ανεκτική σε σχέση με τη βουλγαρική κυβέρνηση και την πολιτική επεξεργασία ε, των αποβλήτων της πρωτεύουσα. Παρά την ανοχή αυτή, οι αρχές δεν άλλαξαν απολύτω τίποτε για να βελτιωθεί η κατάσταση. Πρόκειται για, ένα, για μια χωματερή που είναι ένα βιολογικό όπλο, είναι, πρόκειται για ένα βιολογικό πόλεμο κατά των ε, κατοίκων. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες που εκλείουν διοξίδιο του άνθρακα, θάνη, όπως επίσης και οξύδια ε, θείου και αζότου. Επίσης, ε, ε, προκαλούν πάρα πολλές ασθένειες, όπως για παράδειγμα χάγκρινα. και αυτό οφείλεται κυρίω ε, σε σύγκρουση συμφερόντων στο πλαίσιο τη βουλγαρική κυβέρνηση. Υπάρχουν νέε τεχνολογίε που είναι ήδη διαθέσιμε ε, στην Ευρώπη για την καλύτερη επεξεργασία των αποβλήτων. Όμω οι τεχνολογίε αυτέ οι νέε δεν χρησιμοποιούνται στη Βουλγαρία λόγω αυτών των ε, συμφερόντων και, των, και της διαφθοράς που σας ανέφερα. Όμως δυστυχώς ο, κάθε επίκριση των εμπειρογνωμόνων παραμένει χωρίς απάντηση, παραμένει αναπάντητη και αυτό είναι πολύ επιβλαβές και για τους κατοίκους μας, αλλά και για τις ε, μελλοντικές γενναίες. Είναι επίσης ε, σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές αρχές ε, για την υγεία των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Όσον αφορά τώρα τον κίνδυνο για την υγεία. υπάρχει μεγάλο ποσοστό, υψηλό ποσοστό καρκίνου στην ε, περιοχή. 5 με 6 ε, κρούσματα ε, σκλήρινσης κατά όπως επίσης, και μιλάω για μια πολύ μεγάλη περιοχή της ε, πρωτεύουσας. Εμείς, ως κάτοικοι του Σουχοντόλ ζητούμε με καλύτερη υποστήριξη και μεγαλύτερη πίεση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προ τη βουλγαρική κυβέρνηση, προκειμένου να επιληθεί το πρόβλημα των αποβλήτων του Σουχοντόλ με οικολογικό τρόπο που δεν θα απειλεί τη ζωή των κατοίκων ε, της περιοχής. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω μια συζήτηση εμπειρογνωμόνων, παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είμαι έτοιμο να, ζητήσω να δώσω περισσότερα στοιχεία εμπειρογνωμοσύνη και ευχαρίστω ε, να απαντήσω και σε ερωτήσει σα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να αναφερθώ μία ακόμη φορά στις οδηγίες που δεν έγιναν σεβαστές περί ανακύκλωσης 2001-67. Μπορείτε να τις βρείτε και στα έγγραφα που έχετε στη διάθεσή σας, όπως επίσης και περί άνθρακα 87 του 2003 της Ευρωπαϊκής ε, ε Κοινότητας η έλλειψη συστήματος επεξεργασίας αποβλήτων, η καθυστέρηση και η σύγκρουση πολιτικών συμφερόντων, όλο και περισσότερο βεβαίως δημιουργούν προβλήματα και αυξάνουν τον αριθμό των θυμάτων. Γι' αυτό το λόγο απευθυνόμαστε σε εσά ως τελευταίο μας ε, καταφύγιο. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Ιβανόφ. with regard όσον αφορά, όσον αφορά την διάθεση των απορριμμάτων στην ε, ε, Βουλγαρία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει μία διαδικασία ε, λόγω της παραβιάσεως της σχετικής οδηγίας του 2006 όσον αφορά την διάθεση των οικιακών αποβλήτων. Το 2007 στείλαμε μία επίσημη ε, ε, ενημέρωση στη Βουλγαρία. Το 2008 απεστάλλει μία αιτιολογημένη ε, γνωμοδότηση στην οποία απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 2009 η ε, Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το θέμα στην ε, Ευρωπαϊκή, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω μη συμμορφώσεως και το 2010 η Βουλγαρία υπέβαλε ε, εις ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα μεγάλο πρόγραμμα ε, και η Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει ε, την βιωσιμότητα του συστήματος αυτό ότι έχει επαρκή ε, δυνατότητα ε, για την υγειονομική ταφή και την χρήση των υποπροϊόντων. Το, θα πρέπει όμως να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Πρέπει ολόκληρο ολόκληρο το πρόγραμμα να θεωρηθεί σαν ενιαίο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί το πρόγραμμα αυτό να συνοπτιστεί σε δύο φάσεις. Η μία να ξεκινήσει αμέσως και η δεύτερη να εφαρμοστεί μόλις θα έχει ε, καλυφθεί και η επιπρόσθετη ανάλυση. Έχουμε λοιπόν ενημερώσει τις βουλγαρικές αρχές ότι μπορούν έτσι να ε, εφαρμόσουν ε, ένα πρόγραμμα διαθέσεως από ε, ικανοποιητικό. Όσον αφορά την Σόφια, ως που ε, να κατασκευαστεί και ε, να λειτουργήσει αυτή η εγκατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε επαφή με τις βουλγαρικές αρχές για να εξασφαλίσει ότι το σύστημα διαχείρισης των σχετικών αποβλήτων στη Σόφια ε, θα συνάδει με τις επιταγές της περιβαλλοντολογικές. Ε, μέχρι λοιπόν ε, εφαρμοστεί ε, την, η, η απόφαση αυτή παραμένει η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραπέμψει τη Βουλγαρία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μία συμμόρφωση. Ε, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή διότι δεν έχει εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ε, διάθεση των αποβλήτων. Θέλετε να προσθέσετε κάτι κυρία Πρόεδρε. Στο τέλος καλύτερα. Να δώσω το λόγο στους συναδέλφους καταρχήν. Παρακαλώ. Συνάδελφος Γιατώμα. Благодаря, госпожо председател. Аз ще говоря също на български язик. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω κι εγώ στην Βουλγαρική. Για νιωστή φορά συζητούμε αυτό το ζήτημα στην Επιτροπή μας. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της τελευταίας θητείας ε, το είδαμε. Είναι πράγματι κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό αυτή η αναφορά έχει ημερομηνία 2007 και τώρα είμαστε στο 2011 και αυτό μας δείχνει το ρυθμό των εργασιών της Επιτροπής μας. Ουσιαστικά αυτό είναι μια απάντηση στη συζήτηση που είχαμε για την αποτελεσματικότητά μας. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας δίνει μια επίσημη απάντηση, την έχουμε ακούσει πολλάκις. Μια απάντηση η οποία συμπίπτει με την απάντηση που έλαβα και ως βουλευτής. Σε ερώτηση υποτέθηκε εδώ και κάποιους μήνες. Τίποτα το καινούριο δεν υπάρχει και η κατάσταση που περιγράφεται και που την είδαμε και στην οθόνη, συνεχίζει να είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ρωτήσω το εξή. Ε, πώς ε, φαντάζεται να συνεργαστεί με την κυβέρνηση της Βουλγαρίας μέχρι τη στιγμή που θα κατασκευαστεί το εργοστάσιο επεξεργασίας των μάτων, ε, γιατί μέχρι, τίπο... μέχρι σήμερα τίποτα δεν έχει γίνει για να κατασκευαστεί αυτή η μονάδα και δεν είναι καθόλου σαφή τα πράγματα σε σχέση με τα δύο στάδια. Σε τι συνίσταται αυτά τα δύο στάδια κατασκευής ε, του σταθμού επεξεργασίας αποβλήτων. Ποιες είναι οι πρόσθετες λεπτομέρειες που θα πρέπει να παρουσιαστούν προκειμένου τελικά να εγκριθεί τον λόγο έργο και να κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις. Ε, ποιες είναι οι προθεσμίες που έχει στη διάθεσή τη ο Δήμος της Σόφια για να επιλύσει το πρόβλημα αυτό, γιατί ο πληθυσμός ε, συνεχίζει να ζει σε ένα περιβάλλον που δεν είναι καθόλου υγιεινό. Ποιε πληροφορίες έχουν δώσει λοιπόν οι βουλγαρικές αρχές σε ό,τι αφορά αυτή τη χωματερή στο Σχοντόλ. Βλέπουμε ότι υπάρχει παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ε, η Κομισιόν ε, δεν σκέφτεται να κάνει έναν έλεγχο επιτόπου, γιατί ο πληθυσμός ε, διαμαρτύρεται, απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που φέρνει παρουσία στην απάντησή της, αλλά το ζήτημα παραμένει ακρεμές. Το ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιλήφθη επί του ζητήματος δεν επέφερε κανένα αποτέλεσμα μέχρι σήμερα. Εδώ και τέσσερα χρόνια ήδη επιζητείται λύση στο πρόβλημα αυτό και από ό,τι φαίνεται δεν προκύπτει η λύση. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή και εκτιμώ ότι θα πρέπει να στείλουμε και εμείς ως Επιτροπή μία επιστολή στο Δήμιο της Σόφιας και στην κυβέρνηση της Βουλγαρίας και θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να οργανώσει μια νέα αποστολή ελέγχου στη Σόφια. Ευχαριστώ. Μποστινάρου. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι και κύριοι αναφέροντα. Είναι η ίδια ιστορία. Αναρωτιόμαστε αν υπάρχει δυνατότητα πλέον να αναρωτιόμαστε πόσο καιρό χρειάζεται έχουμε μία αναφορά από το 2007 που δεν έχει ακόμη επιληθεί και είμαστε στις αρχές του 2011. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι προσεκτικά και σοβαρά διερευνά το θέμα της ιδανικής εφαρμογής ενός έργου στο Σχοντόλ. Πολύ ωραία. Αλλά Κύριε πρόσωπε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πριν να κατηγορήσετε την βουλγαρική κυβέρνηση και μπορώ να μαντέψω ποιος ε, ήταν δήμαρχος τότε στη Σόφια. Αλλά δεν είναι σοβαρό τώρα το ερώτημα. Αυτό αστείο είναι τέλος πάντων. Αλλά πέραν των αστεισμών, πείτε μας παρακαλώ κύριε πρόσωπο της Κομισιόν. Πόσο χρόνο χρειάζεστε για να αξιολογήσετε σοβαρά την κατάσταση. Έχετε πληροφορίες τεχνικού χαρακτήρα για τις εξελίξεις εκεί. Έχετε καθόλου πληροφορίες για τον αντίκτυπο αυτής ε, της ε, εγκατάστασης ε, στο περιβάλλον και στη ζωή των κατοίκων. Μάλλον όχι. Κατόπιν, πείτε μας. Αναφερθήκατε σε μία μελέτη Πότε τελικά θα εφαρμοστεί η μελέτη αυτή. Έχετε ένα χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε να μας πείτε ναι αυτή η εγκατάσταση θα αρχίσει να λειτουργεί το Μάρτιο, τον Νοέμβριο, δεν ξέρω πότε. Και μάλλον θα αρχίσει να δημιουργείται το Μάιο τον Νοέμβριο και θα λειτουργεί το 2020. Είναι τμήμα της στρατηγικής του 2020 και ακόμη δεν ξέρουμε τίποτα. Με συγχωρείτε. Αλλά εδώ έρχεστε και μας λέτε κενά λόγια. Δηλαδή έρχεστε εδώ ενώπιον της Επιτροπής μας και τι μας λέτε. Φλερίες, ε, κοιτάξτε εδώ, εδώ δεν μιλάμε για τη βίβλο, ούτε εσείς το Ιερός Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να μας πείτε πότε και πότε η διαδικασία που παραβάση θα είναι αποτελεσματική. Όταν μια κυβέρνηση κράτους μέλους δεν αναλαμβάνει δράση σύμφωνα με την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τελευταίο σχόλιο. Ποιος θα πληρώσει αποζημίωση, τις αποζημιώσεις ε, σε αυτούς τους ανθρώπους ε, που ζουν ε, στην περιοχή και έχει καταστραφεί ζωή τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η βουλγαρική κυβέρνηση, θα πληρώσουν προβλέπονται κάποια κονδύλια, κάποιες αποζημιώσεις που θα δοθούν σε ανθρώπους αυτούς, ε, οι οποίοι χάνουν τις περιουσίες τους και θίγεται η υγεία τους. Πρόεδρε, είναι απολύτως απαραίτητο τελικά να κάνουμε μια συζήτηση και όταν ε, θα εκπονήσουμε αυτήν την έκθεση για τη θήριση των υποβλητών μαζί με την Επιτροπή Περιβάλλοντος να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα για να συζητήσουμε το θέμα γιατί ο τρόπος με τον οποίο απαντούν τα κράτη και διαχειρίζονται το θέμα είναι απολύτως απαράδεκτος. Θα πρέπει... Μάλλον θα πάμε σύντομα στην Βουλγαρία. Τι μήνυμα θα φέρουμε στους βουλγαρούς πολίτες για το νόμιμο αίτημά τους. Τι αξιοπιστία θα έχουμε όταν θα συναντήσουμε τον κόσμο, τους πολίτες. Τίποτα. Γελοί θα είμαστε και εγώ δεν μπορώ να το δεκτώ αυτό. Με συγχωρείτε. Okay. Ε, Ευχαριστώ. Και εγώ συμφωνώ απολύτως με τον Βίτο και νομίζω ότι αυτή η ατμόσφαιρα ατιμορρησίας είναι τώρα ένα πρόβλημα που μας απασχολεί σχετικά με τα σκουπίδια. Δηλαδή παντού θεωρούν ότι είναι αποδεκτό ότι τίποτα δεν συμβαίνει, τίποτα δεν γίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όπου μπορεί να γίνει δεν είναι αδύνατον να επιλύσει κανείς τα προβλήματα των σκουπιδιών και των αποβλήτων και βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι πολύ πιο ισχυρή επ' αυτού. Έπρεπε ήδη εδώ και πολύ καιρό να έχει επιληφθεί και θα έπρεπε επίσης να ζητήσουμε να υπάρξει κάποια συνεργασία ώστε όπου έχουν κάποιο αποτέλεσμα να μπορέσουν να προσφέρουν ιδέες για το πώς θα προχωρήσουμε. Γιατί αν εμείς δεχόμαστε ότι ε, τα απόβλητα είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, δεν αναφέρουμε μόνο στα νέα κράτη-μέλη και στα παλιά επίσης στα παλιά Δεν ε, μας ε, λαμβάνουν στα σοβαρά. Οπότε είναι πολύ άσχημη η κατάσταση και υπάρχουν ε, κραυγαλές αποδείξεις ότι μπορούσαμε να έχουμε επέμβει πριν από χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την, Ευρωπαϊκή, από την Επιτροπή μας εάν συνεργάζεστε με την Επιτροπή στην Κοπεχάγη η οποία ασχολείται με το θέμα αυτό και μπορεί να μας ε, βοηθήσει να αλληλοβοηθηθούμε διότι έτσι όπως έχει κατάσταση τώρα είναι όλα δύσκολα και τα νέα κράτη-μέλη ε, δεν έχουν καθόλου στοιχεία, δεν ξέρουν τι πρέπει να γίνει και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητά άλλο το λόγο. Με συγχωρείτε. Δεν σας είδα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες και να τονίσω ότι τέσσερα χρόνια είναι πραγματικά υπερβολικά και είναι μεγάλη επιβάρυνση για τον λαό που πλήττεται και ε, δεν μπορεί κανείς να καλύψει τα έξοδα υγείας. Αν έχουμε περιπτώσεις καρκίνων, καρκινοπαθών, τι θα γίνει, θα τους πληρώσουμε τις χημειοθεραπείες. Πρέπει να δούμε πόσο σοβαρή η κατάσταση είναι όταν ασθενούν από καρκίνο και θα πρέπει να υπάρξουν πολύ γρήγορες ενέργειες κατά τρόπο ώστε να μειώσουμε ε, τα δεινά των ε, εμπλεκομένων διότι θα έπρεπε μάλλον να κοιτάξουμε πώς θα χειριστούμε καλύτερα την, ε, το θέμα της φύσεως διότι η φύση συμβάλλει πάρα πολύ στην υγεία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Γιάρ. Ε, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε ομάδα αναφορών που αναφέρονται στο θέμα των αποβλήτων και με ενδιαφέρει διότι δεν είναι ότι δεν έχουμε τις τεχνολογίες για να αποφύγουμε αυτές τις καταστάσεις έχουμε ε, μεν ε, τόπους τα φύση των απορριμμάτων αλλά η διαφορά από το μεσαίωνα είναι ότι αντί να είναι στη μέση του δρόμου είναι κάπου παραπέρα. Ε, έχουμε πολλές εναλλακτικέ λύσεις. Ε, είδαμε ότι μπορεί κανείς να τα προστατεύσει και δεν χρειάζεται να μένουν έτσι τα σκουπίδια. Δεν είναι καν θέμα οικονομικό. Δεν είναι ότι υπάρχει στενό της χρημάτων ε, άλλοτε λέγαμε ότι εποχές ε, σοσιαλιστικής ε, υπήρχε κάθε, κάποιος, κάποια χώρο ματερή σε κάθε χωριό. Λοιπόν, όταν ε, ακούω ότι ε, υπάρχουν ε, εκκλήσεις ότι με τα σκουπίδια μπορεί κανείς να κερδίσει χρήματα με τα σκουπίδια ήθελα να το απαντήσω ότι ορισμένοι ναι με το έχουν καταλάβει αλλά από την λάθος κατεύθυνση και εκμεταλλεύονται τα σκουπίδια για να κερδίσουν χρήματα. Λοιπόν, θα έπρεπε ίσως ε, να κάνουμε μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και να δούμε πώς θα διεκπαιρεώσουμε τα θέματα των ε, σκουπιδιών. Ε, διότι βλέπουμε ότι υπάρχουν λογιστικές αξιολογήσεις, μετά υπάρχουν ερωτηματολόγηση, μετά αρχίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απειλεί με δίωξη, αλλά αυτοί που είναι υπεύθυνοι στο το τέλος ε, δεν ε, βλάπτουν μόνο το περιβάλλον αλλά προκαλούν και ε, σωματικές βλάβες, επεμβαίνουν στην υγεία των ανθρώπων και πρέπει να υπάρχει ένας σωστός μηχανισμός εκτός και αν δεν ενδιαφέρεται κανείς. Μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πότε θα ξεκινήσετε πραγματικά. Δηλαδή, πρώτε θα θέσετε τον ακρογωνιαίο λίθο για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε εφαρμόζουμε μία στρατηγική για τα σκουπίδια. Ε, εκτός ε, και αν θα περιμένουμε ε, πάντοτε και πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τις υπάρχουσες χωματερές και με την ε, μετακίνηση ορισμένων ε, που ξεκινούν τώρα. Διότι δεν είμαστε ε, σε αναπτυσσόμενα κράτη, δεν ζούμε πια στο μεσαίωνα, άρα θα έπρεπε κάποια στιγμή τα κράτη-μέλη σωστά και αποτελεσματικά να μπορέσουν να ενδιαφερθούν και να επέφτουν αλλά ξέρω ότι εγώ εκνευρίζομαι. Έχουμε όμως ομάδες, στίβες από αναφορές που ασχολούνται από κλειστικά και μόνο με χωματερές, με τα απόβλητα και ε, δεν βλέπουμε πώς θα υπάρξουν πιο αποτελεσματικά μέσα. Ε, όλοι πιστεύουν ότι ίσως το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να εξοικονομήσουν τα χρήματα αντί να ασχοληθούν με την υγειονομική ταφή. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητά άλλο ε, το λόγο. Ο πρόσωπος της Κομισιόν, όμω ε, ε, μπορείτε να μα πείτε δύο λόγια. Στο τέλο, εσεί θα πάρετε το λόγο αφού απαντήσει η Κομισιόν. Ο πρόσωπος Κομισιόν θέλει να παρουσιάσει τώρα κάποιε απαντήσει. Thank you, Madam Chairman. Uh, Ευχαριστώ πολύ, με Τζόφρι Δεν είμαι ε, Επίτροπος, είμαι τμήματάρχης της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Θα θέλω να απαντήσω στην κυρία Όκεν. Δεν είναι θέμα τιμωρίας, είναι θέμα επίλυσης του ζητήματος. Από την άποψη της τιμωρίας νομίζω ότι κάναμε τη δουλειά μας. Αρχίσαμε διαδικασία επί παραβάση το 2007. Ε, το έτος της προσχώρησης δεν γινόταν νωρίτερα και τώρα αποφασίσαμε να πάμε στο δικαστήριο. Από άποψη λοιπόν ε, επιβολής και ε, ε, δεν ήμασταν οικείς, αλλά αντιθέτω με τη Βουλγαρία. Έχετε δίκιο όμως ότι αυτό που πρέπει να γίνει δεν είναι θέμα να ε, ε, κερδίσουμε πόντους. Το θέμα είναι να λυθεί το πρόβλημα. Και προσπαθούμε στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσής μας ε, να επιλύσουμε το ζήτημα αυτό για να μπορέσει να γίνει ανακύκλωση και επεξεργασία των αποβλήτων. Υπάρχει μια επένδυση 8, 80 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει τα 10 εκατομμύρια και τα υπόλοιπα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν είναι λοιπόν κάτι το οποίο μπορεί κανεί να το κρίνει μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Δεν είμαστε πλήρω ικανοποιημένοι με το πρόγραμμα που υπέβαλαν οι βουλγαρικέ αρχέ. Έχουμε πολλέ επαφέ μαζί του. Ε, πάλι την Παρασκευή θα συναντήσουμε τον αντιπρόεδρο, τον, ε, συγγνώμη, τον υφυπουργό ε, τη περιβάλλοντος και τον αντιδήμαρχο της περιοχής της ε, Βουλγαρίας. Όπως βλέπετε λοιπόν υπάρχουν επαφές με τη βουλγαρική κυβέρνηση. Κάνουμε και επισκέψεις. Οι συναδέλφοί μου από, την αρμόδια, από το αρμόδιο τμήμα της Γενικής Διεθνής Περιβάλλοντος αλλά και από την Επιτροπή Περιφερειών πηγαίνουν συχνά στη Σόφια. Αν λοιπόν καταφέρουμε να έχουμε ε, κάποια προγράμματα σε δύο στάδια, ελπίζουμε μέσα στους ερχόμενους μήνες να υπάρχει μία ε, πρόοδος και σε κάποια χρόνια να υπάρξει οριστική λύση. Ξέρω ότι δεν είναι η καλύτερη δυνατή λύση που μπορεί να δοθεί. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε επαφές με τις βουλγαρικές αρχές και αυτές είναι οι πληροφορίε που μπορώ να σα επιβεβαιώσω ε, για την ώρα. Ευχαριστώ. Ο Ανεφέρον έχει το λόγο για να απαντήσει. Ευχαριστώ. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή όλες τις παρεμβάσεις. Εδώ δεν μιλάμε για χειρώσεις. αλλά ως βουλγαρούς πολίτες ήθελα να σας πω ότι δεν είμαστε και τόσο ανόητοι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η σημερινή κυβέρνηση θέλει να ε, λαμβάνει συγχαρητήρια και ξέρουμε τις ε, ε σχέσεις που υπάρχουν ε, και την, τα παιχνίδια εξουσίας μεταξύ βουλγαρικής κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως είδατε και στην οθόνη τα θύματα. Τελευταία είχαμε το θάνατο ενός 14χρονου κοριτσιού από καρκίνο. Έχουμε θύματα λοιπόν. Αυτό ήθελα να υπογραμμίσω. Και πρέπει να σκηθεί πίεση στην κυβέρνηση. Είπατε ότι δεν είχατε ιδέα. Όμως εμείς ε, ξέρουμε ε, ότι είναι αναρμόδια η δημοσία για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Εμείς πρέπει να ξέρετε ότι δεν εγκρίνουμε αυτό το πρόγραμμα διαχείρισης των αποβλήτων στη Σόφια, γιατί αυτό το έργο θα μολύνει όχι μόνο τη Σόφια, αλλά και όλη τη Βουλγαρία και γι' αυτό είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε σε όλα τα επίπεδα για να έχουμε μία λύση που να σέβεται την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, αλλά ε, κανένας ε, δεν στρέφεται σε εμά γιατί εμείς δεν έχουμε την εξουσία. Κανείς δεν ακούει τους πολίτες. Ενώ έχουμε πάρα πολύ λογικές ιδέες. Αλλά δεν αποτελούμε θμήμα του δίκτυου της διαφοράς, είμαστε από την άλλη πλευρά. Και θέλω να υπενθυμίσω και κάτι άλλο. Το ότι καθυστερεί η επίτευξη λύσης για το πρόβλημα αυτό, αυτό μας εκπλήσει. Αλλά οφείλω να σας πω ότι έχουμε την πρόθεση να προσφύγουμε και στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Η Κομισιόν συνεχίζει να ανέχεται μια πραγματική γενοκτονία από την ε, βουλγαρική κυβέρνηση. Εμείς δεν θα καταλήψουμε στον τον αγώνα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πιστεύω ότι και εδώ Έχουμε ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να επιληθεί. Η Κομισιόν μας είπε ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία, δεν έχει ακόμα ξεκινήσει διαδικασία επί παραβάση ούτε έχει ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία, αλλά είναι σε επαφή με την τοπική αυτοδιοίκηση για να προσπαθήσουν να δώσουν απαντήσεις στα προβλήματα που τίθενται. Συμφωνώ με όλους τους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα αυτής της διαδικασίας. Ε, πιστεύω ότι και εμείς εδώ, σε αυτή την Επιτροπή, θα πρέπει να εργαστούμε, αλλά και η Εκτελεστική Επιτροπή θα πρέπει να εργαστεί επί του ζήτηματος. Αλλά εμείς πρέπει να αισθητοποιήσουμε ότι τα ευρωπαϊκά όργανα, οι ευρωπαϊκές αρχές δεν μπορούν ε, να επιβάλλουν στις τοπικές αρχές πώς θα διαχειριστούν τα τοπικά προβλήματα. Απλώς ε, γίνεται μια παρακολούθηση, μια αποπτία. και επιβάλλονται κυρώσεις ε, στα κράτη. Ε, χρησιμοποιείται το όπλο της μείωσης της χρηματοδότησης. Έτσι λοιπόν ε, είναι σαφές ότι οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται είναι συνεχούς προσοχής ε, και παρακολούθησης. Πιστεύω ότι υπάρχουν πιο μεγάλα προβλήματα που ξεπερνούν το μεμονωμένο ζήτημα του σταθμού ε, της επεξεργασίας των αποβλήτων που δεν έχει εγκριθεί εγκαίρως. Πρέπει να αναλύσουμε αυτά τα ζητήματα και θέλω να επαναλάβω πόση σημασία προσδίδουμε εμείς ως Επιτροπή στην αναγκαιότητα να γίνει μια ολοκληρωτική μελέτη του ζητήματος των αποβλήτων στην Ευρώπη. Γιατί είναι ένα ζήτημα που προκύπτει συνεχώς στις διάφορες χώρες με παρόμοιους τρόπους πολλές φορές. Έτσι λοιπόν η έκθεση που ζητήσουμε και ελπίζω να μπορεί να εγκριθεί από την Προεδρία το συντομότερο Ελπίζω να δεν προς την κατεύθυνση, δηλαδή να αναζητήσει απαντήσεις σε ερωτήσεις που ίσως ακόμη δεν έχουμε θέσει κατά ολοκλήρωση, καθώς συνεχίζουμε να αναλύουμε μονομένες περιπτώσεις και δεν βλέπουμε το σύνολο του προβλήματος, τη συνολική εικόνα. Η Προεδρία όμως δεσμεύεται να προσπαθήσει να επιταχύνει τις διαδικασίες εξέτασης ε, αυτής της αναφοράς ε, για το θέμα των αποβλήτων. Τώρα για την ίδια την αναφορά ε, φυσικά θα τη διατηρήσουμε ανοιχτή και περιμένουμε η Εκκληστική Επιτροπή να επιταχύνει τις διαδικασίες αυτού του διοργανικού έργου και ακόμη και σε αυτή την περίπτωση τα μέλη της Επιτροπής ε, θεωρούν ότι είναι χρήσιμο η Επιτροπή Αναφορών να στείλει ένα σημείο με μια επιστολή στις τοπικές αρχές προκειμένου να έχουμε περαιτέρω ανατροφοδότηση και για να επιταχύνουμε περισσότερο την εξέβρεση λύσης. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι θεωρούν ότι είναι χρήσιμο να στείλουμε μια επιστολή στις αρμόδιες αρχές. Δεν ξέρω, αυτό το είπαμε και πριν. Πιστεύω ότι γνωρίζετε, το είχαμε και στις ανακοινώσεις του φακελού, ότι εμείς ήδη έχουμε στείλει μια επιστολή, αλλά δεν λάβαμε καμία απάντηση. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι ήταν χρήσιμο να ξαναγράψουμε την επιστολή και πιο έντονα να ζητήσουμε μια απάντηση στις προβληματικές που τίθενται. Ε, ευχαριστώ τον αναφέροντα και περνώ στο επόμενο σημείο. Έχουμε την αναφορά 78-2007 στο σημείο 9, εδώ είναι παρόν και ο αναφέρον, ο κύριος Βορίδης και θα του δώσω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συγκεκριμένη υπόθεση ξεκινάει με την ψήφιση του νόμου 3164 του 2003 με την οποία ολοκληρώνω το Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείριση Θερών Αποβλήτων τη Περιφέρεια Αττική. Με αυτόν τον νόμο ορίστηκαν ω θέσει εγκατάσταση ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων, δύο θέσει μεταξύ άλλων, η θέση Μαύρου Βουνό Γραμματικού και η θέση Βραγώνη Κερατέ Λαμπριωτική. Θα ήθελα απλώ να τονίσω ότι στο συγκεκριμένο νόμο, στην παράγραφο 2, ορίζεται ότι θα έπρεπε να φτιαχτούν ακόμα έξι θέσει κεντρικών σταθμών μεταφόρτωση αποβλήτων στην περιφέρεια Αττικής. Το λέω αυτό και κρατήστε το στην σκέψη σας, διότι το βασικό επιχείρημα το οποίο θα αναπτύξω εδώ είναι ότι στην πραγματικότητα η ελληνική διοίκηση δεν προχωρά σε ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, αλλά στην πραγματικότητα εγκαθιστά χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, χωρίς να έχει κάνει ό,τι πρέπει, όπως ορίζει η σχετική κοινοτική οδηγία, για να μειώσει τον συνολικό όγκο των βιοαποδομήσεων αποβλήτων ώστε να περιορίζεται ο όγκος των αποκλήτων τα οποία θα προχωρούν σε υγειονομική ταφή. Μετά τον νόμο αυτό, τον νόμο του 2003, υπήρξαν δύο αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτούσε την κατασκευή χώρων χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στις δύο συγκεκριμένες θέσεις. Οι αποφάσεις αυτές ήταν η 5509, η οποία εγκρίθηκε στις 21 Δεκάτου του 2004, και η 55 ε, και η 2004-16C ε, η οποία αφορούσε την ε, κερατέα. Μέσα στις αποφάσεις αυτές υπήρξαν έξι ειδικοί όροι, περιλήφθηκαν έξι ειδικοί όροι. Ο όρος 6 έλεγε ότι σε περίπτωση μη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων ή των ανωτέρων υποχρεώσεων, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε την υποχρέωση να σταματήσει την χρηματοδότηση του έργου, να προχωρήσει στην άρση χρηματοδότηση του έργου. Εγώ εκείνο το οποίο ισχυρίζομαι είναι ότι ουσιαστικά κανένα από του πέντε όρου που έθετε η συγκεκριμένη απόφαση, οι συγκεκριμένε δύο αποφάσει για την χρηματοδότηση των έργων δεν έχουν τηρηθεί. Καταρχά είναι προφανέ ότι δεν έχει τηρηθεί κανένα χρονοδιάγραμμα. Και δεν έχει τηρηθεί κανένα χρονοδιάγραμμα γιατί σύμφωνα με τι αρχικέ αποφάσει θα έπρεπε η ημερομηνία περάτωση των έργων να είναι το 2007, ενώ κανένα από τα δύο έργα δεν έχει περατωθεί μέχρι σήμερα. Η ημερομηνία έναρξης των έργων έπρεπε να είναι το 2005. Τα έργα, το έργο στο γραμματικό ξεκίνησε αρχές του 2009, ενώ υπάρχει ένας ισχυρισμός, τον οποίο θα ακούσετε από την πλευρά της ελληνικής διοικήσεως, ότι δήθεν το έργο στην ε, Κερατέα ξεκίνησε στις 10 του του 2010. Κρατήστε αυτή την ημερομηνία γιατί υπήρξε μια παράταση, κατά τη γνώμη μου κακός, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτέλεση του έργου μέχρι 31 του 2010. Στα κείμενα τα οποία σας έχει διανύμει στην απάντησή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρίζεται ότι δεν ήταν δυνατόν να ξεκινήσουν τα έργα διότι υπήρχαν δικαστικές εμπλοκές. Αυτό είναι εντελώ ανακριβέ. Δικαστικέ εκκρεμότητε βεβαίω και υπήρχαν, ουδέποτε όμω χορηγήθηκε οποιαδήποτε αναστολή εργασιών από το Συμβούλιο τη Επικρατεία. Καθόλου το χρονικό αυτό διάστημα, εάν ήθελε, η ελληνική δίκηση μπορούσε να είχε ξεκινήσει και εκτελέσει τα έργα. Η πραγματικότητα όμω είναι ότι η ελληνική δίκηση όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν προχωρούσε σε οποιαδήποτε εκτέλεση των έργων για τον απλούστατο λόγο ότι δεν είχε επιλέξει την τεχνολογία διαχείρισης των απορριμμάτων, δεν είχε αποφασίσει να χρηματοδοτήσει την κατασκευή εργοστασίων, τα οποία έπρεπε να χρηματοδοτήσει με δικά της χρήματα, προκειμένου να υπάρχει προεπεξεργασία των απορριμμάτων και να μην αναποτίθενται εκεί ανεπεξέργαστα απορρίμματα και επομένως εντελώς εκδικού της φάλματος, εκδικής της ολιγορίας και εκδικής της αμελίας, έχει ε, καθυστερήσει και όχι μόνο έχει καθυστερήσει, αλλά σήμερα δεν διαφυλάσσονται κάνει βασικέ προποθέσει για τη διαχείριση των απορριμμάτων, που είναι να έχει προπάρξει ε, επεξεργασία των απορριμμάτων. Στον όρο 2 τη συγκεκριμένη αποφάσεω, αναλαμβάνουν την υποχρέωση η ελληνική δίκηση να διασβαλίσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι δήμοι που θα εξυπηρετούνται από τα συγκεκριμένα έργα θα έχουν επιλέξει συστήματα προεπεξεργασία πριν τη διάθεσή του σε χώρο υγειονομικής ταφή, δηλαδή διαλογή, ανακύκλωση των μη οργανικών αποβλήτων που θα αποσκοπούν στο να μειωθεί ο όγκο ή η επικινδυνότητα των αποβλήτων. Εγώ λοιπόν ακόμα και τώρα θέτω το ζήτημα ότι μέχρι σήμερα οι Δήμοι, επειδή αντιτίθενται στην δημιουργία αυτών των χώρων υγειονομική ταφή, δεν έχουν επιλέξει κανένα τέτοιο σύστημα. Επομένω είναι προφανέ ότι ο συγκεκριμένο όρο 2 δεν εκπληρώνεται. Ο όρο 3 τη εγκριτική απόφαση λέει ότι θα έχει, πρέπει να έχει υπάρξει μία μείωση ύψου 25% θα έπρεπε να έχει επιτευχθεί μέχρι το 2009 μείωση 25% σε σχέση με την ποσότητα των βιοαπικοδομήσιμων αστικών υποβλήτων στην Ελλάδα. Ο όρο αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει εκπληρωθεί. Θα έπρεπε επίση, πριν την τελική πληρωμή βεβαίω, σύμφωνα με τον όρο 5, να έχουν υπάρξει υποδομέ, δηλαδή να έχει τεθεί σε ενέργεια το σύστημα προεπεξεργασία πριν τη διάθεσή του σε χώρο υγειονομική ταφή, διαλογή και ανακύκλωση των μη οργανικών υποβλήτων, καθώ και το σύστημα συλλογή των ειδικών αποβλήτων, είναι προφανέ ότι τα συστήματα αυτά δεν βρίσκονται ακόμα σε λειτουργία. Η αντίρρησή μα, λοιπόν, ε, κυρία Πρόεδρε, σε σχέση με τι συγκεκριμένε αποφάσει είναι, πρώτον, ότι υπάρχει μια διαρκή παράταση των προθεσμιών, η οποία στην πραγματικότητα διευκολύνει την ελληνική δίκηση στο να μην συμμορφώνεται με τι υποχρώσει που θέτει η Επιτροπή. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διαρκή παράταση των προθεσμιών. Δεύτερο, Υπάρχει μία ακόμα υποχρέωση ότι θα έπρεπε οι ανεξέλεγκτοι χώροι υγειονομική ταφή, η ΧΑΔΑ, θα έπρεπε να έχουν κλείσει και αυτοί οι χώροι είναι ακόμα εν λειτουργία. Επομένω, καμία από τι προποθέσει που η ίδια η εγκριτική απόφαση τη Επιτροπή θέτει για την χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων δεν έχει εκπληρωθεί. Αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί νέα εμπλοκή στο θέμα τη υποθέσεω τη κερατέα, διότι υπάρχει απόφαση του Ειρηνοδικίου Λαβρίου, την οποία θα τη δώσω να αναγνωριστεί στο σχετικό, με την οποία απαγορεύεται η συνέχιση των έργων, ακούστε όμως γιατί, μέχρι να συντελεστεί αναγκαστική απαλωτρίωση. Δηλαδή, από το 2004 που υπάρχει σε εξέλιξη το συγκεκριμένο έργο, η ελληνική διοίκηση δεν έχει κάνει τις απαλωτριώσεις στην Κυρατέα. Να εκπονηθούν μελέτες που προβλέπονται από την Εργολαβική Σύμβαση. Δεν έχουν ακόμη εκπονήσει τις μελέτες και δεν μπορούσαν να τις προσκομίσουν στο δικαστήριο. Να αποφανθούν οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες περί της μη υπάρξης αρχαιολογικών ευρημάτων στο χώρο αυτό. Δεν έχει υπάρξει τέτοια απόμφαση. Και τέλο, να εκδοθούν σχετικέ πολεοδομικέ άδειε. Δεν έχουν καταφέρει ακόμα ούτε τι πολεοδομικέ άδειε να εκδώσουν. Το λέω λοιπόν αυτό, διότι είναι προφανέ ότι με την λειτουργία και με τον τρόπο αυτόν με τον οποίο αντιμετωπίζει η ελληνική δίκηση το θέμα και των δύο συγκεκριμένων χώρων υγειονομική ταφή, αλλά και εν γέννη την διαχείριση των απορριμμάτων, δεν διασφαλίζονται τα βασικά που θέτουν οι εγκριτικέ αποφάσει. Απορώ δε γιατί η Επιτροπή δεν έχει επιβάλει όσα θα έπρεπε να επιβάλει, που είναι κυρίω η άρση τη χρηματοδότηση των δύο έργων. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε. Ζανκρέμις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you, Madam Chairman. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η διαφορά της ε, υπόθεση αυτή σε σχέση με, με τις προηγούμενες είναι ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχει αντίδραση των κατοίκων ε, σε σχέση με δύο προγράμματα που θα λύσουν το πρόβλημα. Δηλαδή, οι δύο χώροι υγειονομική ταφής ε, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να οδηγήσουν στο κλείσιμο των παράνομων χωματερών ε, στις οποίε αναφέρθηκε ο κύριος Βορύδη. και στην περιοχή υπάρχουν πάνω από πέντε παράνομες χωματερέ για τις οποίες καταδικάστηκε η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επομένως, ε, η κατασκευή των χώρων υγειονομικής ταβής ε, ακόμη και στο πλαίσιο των όρων που ανέφερε ο κύριος Βορύδης είναι η λύση για το κλείσιμο των παράνομων χωματερών που υπάρχουν στην περιοχή, που ρηπαίνουν το περιβάλλον και που είναι βέβαια απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Η περίεργη κατάσταση με τα δύο αυτά προγράμματα είναι ότι θα έπρεπε να είχαν ε, αρχίσει διαφορετικά με ολοκληρωμένες διαχειρήσεις επεξεργασίας αποβλήτων, δηλαδή με διαλογή, κομποστοποίηση, ε, με δυνατότητα ανάκτηση ενέργειας κλπ. Αυτό έχει προγραμματιστεί να γίνει. Όπως... Διότι η ιδέα είναι να υπάρξει αυτή η ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων και στις δύο περιοχές και θα υπάρξουν και διαγωνισμοί υπό την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και ε, ελπίζουμε να συγχρηματοδοτηθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, απαντώντας ε, στην γενική σας ανησυχία, κυρία Πρόεδρε, ότι θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη τα προβλήματα Τη διαχείριση αποβλήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα έλεγα το εξή, ότι τώρα που έχουμε αυτή τη νέα οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα και που άρχισε να ισχύει από την 12η Δεκεμβρίου του 2010, τα δύο βασικά προβλήματα είναι η χωροταξία και η χρήση της γης από τη μία και η κοινωνική αποδοχή από την άλλη. Διότι αν δεν υπάρχει ούτε η χωροταξία ε, για την χρήση της γης... Ε, αν υπάρχουν λοιπόν προβλήματα ε, είτε σε τοπικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο και δεν γίνονται σεβαστοί οι διάφοροι όροι στα διάφορα επίπεδα, σαφώ υπάρχει και κοινωνική αντίσταση. Τώρα, η ιδιαιτερότητα τη ελληνική περίπτωση, αν μπορώ να την αποκαλέσω έτσι, είναι ότι οι πολίτε γνώριζαν από την αρχή, από τη δεκαετία του 90, ότι στι δύο αυτέ περιοχέ θα, θα υπήρχαν εγκαταστάσει διαχείριση αποβλήτων. Δυστυχώ όσο περισσότερο καθυστερεί η διαδικασία, τόσο η κοινωνική αποδοχή γίνεται δυσκολότερη. Γιατί οι κάτοικοι έχουν βεβαίως ε, περιουσίες, έχουν ε, ε, ιδιοκτησία, έχουν αυτό το σύνδρομο να μην γίνει στην πλάτη μου κάτι και πρέπει να πω βέβαια ότι αυτή η αδράνεια κάπως δημιουργεί προσδοκίες κιόλα για τους ε, κατοίκους ότι οι εγκαταστάσεις που είχαν προβλεφθεί και προγραμματιστεί δεν θα κατασκευαστούν ποτέ και ότι συνεπώς μπορούν να συνεχίσουν ε, να ε, έχουν την ιδιοκτησία τους χωρίς να υπάρξουν εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων στην περιοχή τους. Τώρα λοιπόν που έχουμε αυτήν τη νέα οδηγία που κωδικοποιεί τις καλύτερες τεχνολογίες, καλύτερες δυνατές τεχνολογίες και υπάρχουν και κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ανέφερε και κάποιος άλλος συναδελφός σας, νομίζω ότι θα έπρεπε να υπερβούμε αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και έχει δίκιο ο κύριο Βορύδη όταν λέει ότι υπήρξαν πολλέ καθυστερήσει στην εφαρμογή ενός ε, μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείριση αποβλήτων. Αλλά από κάπου πρέπει να αρχίσει κανεί. Γιατί Αν δεν, αν δεν, κατασταθούν, αν δεν ε, κατασκευαστούν οι ε, χώροι υγειονομική ε, ταφή, είτε στο γραμματικό που έχει ήδη ξεκινήσει και είναι γεγονό ότι στην Κερατέα υπάρχουν κάποια προβλήματα και ότι όντως υπήρξε κάποια απόφαση δικαστηρίου να καθυστερήσει η έναρξη της διαδικασίας, αλλά όταν έφτασαν οι προσφυγές στο ανώτατο δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο δεν ε, διέταξε την αναστολή των ε, εργασιών και θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι υπάρχουν τρεις αποφάσεις ε, δικαστηρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας που επιβεβαιώνουν το που θα λάβουν χώρα ε, τα προγράμματα και απορρίπτουν όλη την επιχειρηματολογία που παρουσίασαν ε, ε, οι κάτοικοι και η περίπτωση επί της οποίας επιλήφθηκε το δικαστήριο, το πρωτοδικείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ότι θα υπάρξει ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση αλλά και αυτό απορρίφθηκε. Επομένως, όσον αφορά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει παράβαση της νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να διαπιστωθεί κάτι τέτοιο και επιπλέον ε, το ανώτατο δικαστήριο στη συγκεκριμένη χώρα ε, αποφάνθηκε, είπε ότι μπορεί να συνεχίσει ε, η κατασκευή του έργου. Είναι γεγονός ότι υπάρχει βέβαια ιδιαίτερη αντίσταση και υπάρχουν και κάποιοι όροι οποίοι όντως πρέπει να πληρούνται, πρέπει να γίνει πολλή δουλειά. Όμως ε, οι προσδοκίες είναι ότι θα αρχίσουν σύντομα οι εργασίες, αυτό τουλάχιστον μας είπε η ελληνική κυβέρνηση και αν δεν γίνει κάτι τέτοιο δεν θα γίνει και η Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει συγκατατεθεί, ούτε έχει δώσει ούτε λεπτό του ευρώ ε, για ε, τους χώρους υγειονομικής ταφής της Κερατέας. Έχουμε δώσει μία προκαταβολή ε, για το γραμματικό που έχουν ξεκινήσει τα έργα και συνεχίζουν κανονικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαλαβράκος, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Εν ώψη του γεγονότο ότι στην ατζέντα της Επιτροπής μας είχε εγγραφεί το θέμα αυτό, ε, την περασμένη εβδομάδα επισκέφθηκα τους χώρους ε, ε όχι του γραμματικού της Κερατέας. Ε, τη στιγμή που μιλάμε και σε ένα χρονικό διάστημα 20 έως 30 ημερών περίπου η περιοχή αυτή είναι ανάστατη έχουν εγκατασταθεί δυνάμεις αστυνομικές και από την άλλη πλευρά υπάρχει η τοπική αυτοδιοίκηση, όλοι οι δήμαρχοι της περιοχής και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι αρνούνται να υιοθετήσουν την εξέλιξη αυτού του έργου το οποίο δεν έχει αρχίσει καθόλου βεβαίω. Από την έρευνα που έκανα διαπίστωσα το εξή και βεβαιώθηκε από αυτά τα οποία είπε και ο κύριος εκπρόσωπος της Επιτροπής. Πρώτον, η οικονομική υποστήριξη του έργου δεν υπάρχει. Επομένως υπάρχει κίνδυνος να αρχίσει ένα έργο το οποίο θα εξελιχθεί σε παράνομη και αυτό και να προσθεθεί στις πέντε υπάρχουσες παράνομες χωματερές στην περιοχή άλλη μία. Δεύτερον, δεν υπάρχουν ακόμη τα χρήματα, δεν έχουν δοθεί ακόμη τα χρήματα για να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες των περιοχών στους οποίους θέλει να εγκατασταθεί ή κατά το σχέδιο, κατά τις σχεδίες της κεντρικής κυβέρνησης, η χωματερή της Κερατέας. Και τρίτο και το σπουδαιότερο, όπως σας σήμερα ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, από τη δεκαετία του 90 συζητιέται η εγκατάσταση χωματερής στην περιοχή εκείνη. Την ίδια περιοχή η κεντρική κυβέρνηση επέτρεψε το διπλασιασμό των κατοίκων της περιοχής. Ακριβώς η περιοχή εκείνη έχει τη μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού στο λεκανοπέδιο της Αττικής από το 2003 και μετά εν ώψη μάλιστα του γεγονότος ότι γυτνιάζει με το, η Κερατέα με το κεντρικό αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος όπου η ε, σώρευση του πληθυσμού την τελευταία οκταετία είναι περίπου κατά 60% μεγαλύτερη. Συνεπώς τα δεδομένα υπό τα οποία σχεδιάστηκε η χωματερία αυτή έχουν ανατραπεί στο σύνολό του. Από την άλλη πλευρά δεν φαίνεται ότι είναι έτοιμη η ελληνική κυβέρνηση τόσο οικονομικά αλλά όσο και από πλευράς σχεδιάσεως των λεπτομεριών της εγκαταστάσεως να υποστηρίξει μια ταχεία διαδικασία εις τρόπον ώστε οι άνθρωποι αυτοί της περιοχής και να αποζημιωθούν αλλά και να έχουν μια σύγχρονη χωματερή. Υπό τα δεδομένα αυτά πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι δυνατή η συνέχιση του, της κεντρικής σχεδιάσεως της κυβέρνησης, της ελληνικής, για χωματερή στην περιοχή εκείνη και πιστεύω ο Τσινάμα ότι πρέπει να εκτιμήσουμε ιδιαίτερο το γεγονός ότι υπάρχει πολύ έντονη κοινωνική αναταραχή η οποία εν ώψη και της οικονομικής κρίσης που υπάρχει στην Ελλάδα μπορεί να εγκυμονεί ευρύτερους κινδύνους από ό,τι υπολογίζουν οι κάποιοι της κυβέρνησης της ελληνικής. Και δεν ξέρω μια θριαλίδα τι μπορεί να οδηγήσει, τι μπορεί να οδηγήσει την ε, περιοχή και ιδιαίτερα το νεκαρομέδιο της Αττικής το οποίο είναι το πολυπιθέστερο και έχει κατοίκους οι οποίοι κυρίως πλήττονται από την οικονομική κρίση διότι είναι εργαζόμενοι οι οποίοι απελήθησαν, δημόσιοι υπάλληλοι των οποίων μοιάθησαν οι αποδοχές κατά τρομερά ποσοστά και εν πάση περιπτώσει η, η όσμωσή μου είναι ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται στα όρια της αυτή τη στιγμή, το οποίο πρέπει να το συνεκτιμήσουμε εμείς σαν Επιτροπή. Επιπλέον θα ήθελα να πω το εξή ότι ε, από την ε, εμπειρία μου πολιτικού είναι ότι ε, οι πολιτικοί πολλές φορές θεωρούμε ότι κρινόμαστε από τους λόγους μας. Δεν κρινόμαστε από τους λόγους μας, κρινόμαστε από τα έργα μας. Και το δεύτερο είναι ότι πιστεύουμε ότι έχουμε απεριόριστο χρόνο. Δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο πιστεύω ότι πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα στην περιοχή της Κερατέας και να δημιουργήσουμε έντονη αντίδραση προς την ελληνική κυβέρνηση η οποία πάει στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα προκαλώντας την κοινωνική ανοχή των κατοίκων της περιοχής χωρίς να έχει ουσιαστικό σχέδιο. Πράγμα το οποίο βεβαιώθηκε και από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Non ci sono... Ε, Ευχαριστώ. Ε, εγώ ε, σκέφτομαι ένα, μια σύγκριση με άλλα θέματα δηλαδή ε, το θέμα του χρονοδιαγράμματος και εδώ πάμε στο 2007 πίσω οπότε και σε αυτό συμφωνώ με τον συνάδελφο που μόλις μίλησε απάντησε από την Επιτροπή λίγο γιατί τελειώνει η συζήτηση αυτή αυτό που ήθελα να σας πω είναι το εξής. Ουσιαστικά υπήρξαν ε, καθυστερήσεις και υπάρχει τίμημα των καθυστερήσεων, ότι δηλαδή έχει αυξηθεί η κοινωνική αντίδραση και όπως άλλωστε ανέφερε ο κύριος Αλαβράκος, έχει διπλασιαστεί ο πληθυσμός της περιοχής αυτής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο αυξάνεται η αντίδραση υπό αυτές τις προϋποθέσεις και ποια είναι η ποσότητα αποβλήτων που παράγεται, την οποία θα πρέπει να διαχειριστούμε σύμφωνα με ε, την ε, κοινοτική ε, θεσία. και από την δεκαετία του 90 στην Αττική έχουμε μόνο τρεις χώρους όπου μπορεί να υπάρχει διαχείριση αποβλήτων. Λοιπόν, ο συνδυασμός της κοινωνικής αντίδρασης και της διαγραφής αυτής της λύσεως είναι ότι οι άλλοι δύο χώροι θα χρειαστεί να χειριστούν περισσότερα απόβλητα σε, ε, κάπου όπου έχει διπλασιαστεί η παραγωγή αποβλήτων και στην Κερατέα υπάρχει κοινωνική αντίδραση και λυπούμεθα πάρα πολύ που σημαίνει αυτό και υπάρχει και μία παράνομη χωματερή. Άρα ο υπεύθυνο για να κλείσει την παράνομη χωματερή αντιδρά στην δημιουργία της νέας χωματερής σύμφωνα με τις αρχές ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ο κύριος Βορύδης από ό,τι αντιλαμβάνουμε δεν αντιδρά στην δημιουργία της χωματερής αλλά στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει το πρόγραμμα αυτής της υγειονομικής ταφής. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από κάπου. Και αυτό άλλωστε το συζητήσαμε και προηγουμένως στην περίπτωση της Σόφιας. Μία πρώτη γεωνομική ταφή είναι μία λύση διότι θα μπορέσει να δεχτεί ε, τα απορρίμματα που μέχρι στιγμής οδεύουν στην παράνομη χωματερή και συγχρόνως θα μπορέσετε να δημιουργήσετε και τις επιπλέον εγκαταστάσεις. Υπάρχει μία απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου αν όλα πάνε καλά προβλέπονται εκατομμύρια για τη δημιουργία αυτής της υγειονομική ταφή, Μέχρι στιγμής δεν έχει καταβληθεί τίποτα, αλλά όπως είπα θα παρακολουθήσουμε και αν δούμε ότι δεν ξεκινεί η εργασία ή υπάρχουν καθυστερήσεις θα ε, καθυστερήσουμε κι εμείς ή θα μειώσουμε τη χρηματοδότηση και αν θέλει η Ελλάδα να προχωρήσει θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει ε, εθνικούς πόρους. Αλλά υπάρχει ένας ε, φαύλος κύκλος όπου βλέπετε ότι οι κρίκοι μίας αλυσίδα συνδέονται και τώρα η λύση είναι η δημιουργία της, του χώρου υγειονομικής ταφής. Ευχαριστώ. Και τώρα ο Ετών έχει ένα λεπτό για να απαντήσει. προφανώς nothing has been paid because nothing has been done. Κοιτάξτε, δεν έχει καταβληθεί τίποτα γιατί τίποτα δεν έχει γίνει. Κα, δεν έχει καταβληθεί τίποτε. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να πω δύο πράγματα μόνο σχετικά με την έννοια της κοινωνικής αποδοχής ή της κοινωνικής αντίθεσης και θα πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία σε κάθε μέτρο η οικοδόμηση της κοινωνικής συνένεσης να συνδέεται με μια, αν θέλετε, παράλληλη στρατηγική που ακριβώς οδηγεί, οδηγεί στην ομιμοποίηση. Τι θέλω να πω με αυτό. Όταν λοιπόν έχει υπάρξει ένας νόμος το 2003 και σήμερα βρισκόμαστε το 2011, θα έπρεπε με βάση την οδηγία του 1999 η Ελλάδα να έχει μειώσει κατά 50% τα πρώτα 8 χρόνια από το 1999, δηλαδή μέχρι το 2007, τον όγκο των βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην υπήρχε ανάγκη για έναν τέτοιο σχεδιασμό, μπορεί να μην υπήρχε ανάγκη να φτιαχτούν δύο καινούργιοι χώροι υγειονομικής ταφής, εάν είχαν ακολουθεί, ακολουθηθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα διαφορετικές πολιτικές. Πώς λοιπόν σήμερα θα οικοδομηθεί κοινωνική συνένεση όταν οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η κυβέρνηση κάνει το πιο απλό πράγμα, δηλαδή φτιάχνει έναν χώρο υγειονομική ταφή, για να πάει να θάψει εκεί απορρίμματα, μη ακολουθώντα όλη αυτή την πολιτική και τη στρατηγική που έπρεπε να ακολουθηθεί και που υποδεικνύουν σειρά οδηγιών τη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι που μα δημιουργεί εντύπωση από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι σε τελευταία ανάλυση η εγκριτική απόφαση είναι ένα νομικό κείμενο. Η εγκριτική απόφαση έχει προποθέσει. Όταν δεν εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις αυτές, σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση κάτι δεν έκανε καλά. Γιατί πρέπει να επιβραβεύεται με τη χρηματοδότηση την στιγμή που ακριβώς κάτι δεν έκανε καλά. Αυτή είναι η δική μας θέση. Ομολογώ ότι δεν κατανοώ ποια είναι η θέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά μία τελευταία κουβέντα. Σε ό,τι αφορά τους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, αυτό είναι επίσης απολύτω ανακριβές και είμαι βέβαιος ότι αποτελεί προϊόν παραπληροφόρηση τη ελληνική διοίκηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι χώροι ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων στην περιοχή υπάρχουν γιατί οι συγκεκριμένοι δήμοι δεν γίνονται δεκτοί στον νέο σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής που έχει την διαχείριση των απορριμμάτων. Δεν του δέχονται τα απορρίμματά του στι ήδη νομίμω λειτουργούσε εγκαταστάσει. Αυτό με απόφαση του νέου συνδέσμου Δήμου και Κοινοτήτων Νομού Αττικής. Όχι γιατί οι ίδιοι οι Δήμοι δεν θέλουν να αποθέσουν τα απορρίμματά του, εκεί που υπάρχουν νόμιμοι χώροι υγειονομική ταφή και ταυτοχρόνω και τεχνικέ επεξεργασίε των απορριμμάτων. Εγώ εκείνο λοιπόν το οποίο λέω είναι ότι δεν είναι δυνατόν οι κάτοικοι να υποστούν την επιβάρυνση του περιβάλλοντο, την καταστροφή αρχαιολογικών μνημείων, την στιγμή ακριβώ που δεν έχουν υπάρξει συνολικά μέτρα για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτό είναι που το οδηγεί, σε έλλειψη δικαιώσεω των πολιτικών και αυτό είναι που δημιουργεί το μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, επαναλήφθηκε το πρόβλημα. Έχουμε εδώ ένα χρονοδιαγράμμα που δεν σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών. Έτσι, λοιπόν, βάσει και της πρότασης του συναδελφού Μποστινάρου θα σκεφτούμε να συνομιλήσουμε με τον ε, κύριο Σουφκόβιτς για να βελτιώσουμε τις ε, διοργανικές επαφές. Νομίζω ότι είναι μια χρήσιμη πρόταση αυτή και στην περίπτωση αυτή έχουμε δυσκολία συσχέτισης με τις τοπικές αρχές που δεν σέβονται τα χρονοδιαγράμματα αλλά ούτε και τους τρόπους ε, δράσης και Εδώ θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ και με τους συναδέλφους που πήραν το λόγο, γιατί ε, και εξακολουθούμε να περιμένουμε μία απάντηση από τις τοπικές αρχές που θα έπρεπε να αναφέρεται στην διαδρομή που θα έπρεπε να ακολουθηθεί και που έχει επιλεχθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή. Έτσι λοιπόν υπάρχει πρόβλημα και με την Κομισιόν. Ε, έχουμε λοιπόν ε, μία αναφορά που ε, δυστυχώς θα πρέπει να παραμείνει ακόμα ανοιχτή, το λέω το δυστυχώς λόγω των συνεπειών που προκύπτουν και θα πρέπει εμείς να παρακολουθούμε στενά αυτές τις υποθέσεις και φυσικά να ζητήσουμε και feedback από τις τοπικές ευχές και από την Εκτελεστική Επιτροπή. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο, στην επόμενη αναφορά. Είναι εδώ ο συνάδελφος Ιμπράσας. La parola Ο κύριος Ιμπράσας έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα μίλησαμε πάρα πολύ για το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων η δική μου αναφορά επίσης έχει να κάνει με τη διαχείριση των αποβλήτων, αλλά όχι με τους χώρους υγειονομικής ταφής, αλλά με την αποτέφρωση των αποβλήτων. Ξέρω ότι δεν είναι προτεραιότητα αυτό το θέμα, αλλά αποτελεί επίσης τμήμα της επεξεργασίας αποβλήτων. Είναι δυνατόν να έχουμε αποτέφρωση αποβλήτων. Η δική μου αναφορά έχει παρουσιαστεί. Να σας πω ότι εγώ δεν είμαι μόνο αναφέρον, αλλά είμαι και ευρωβουλευτής. Και γιατί αποφάσισα να παρουσιάσω αυτή την αναφορά. Μία συγκεκριμένη επιχείρηση στο Βίλνιους, μια αρκετά μεγάλη εταιρεία, συμμετέχει σε πάρα πολλές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και τώρα θέλει να προβεί στην αποτέφρωση αποβλήτων. Έχει ένα αγροτεμάχιο και αποφάσισε εκεί να οικοδομήσει μια μονάδα αποτέφρωσης των αποβλήτων, όμως ε, αυτό το κομμάτι βρίσκεται στην δυτική πλευρά, πάρα πολύ κοντά σε ε, κατοικήσιμες ε, περιοχές του Βίλνιους. Εκεί βρίσκεται περίπου το 30% του πληθυσμού της πόλης. Επίσης, ε, αυτή η τοποθεσία βρίσκεται κοντά σε προστατευόμενες ε, περιοχές που θα συμπεριληφθούν στο δίκτυο Natura 2000. Ακόμη, υπάρχει ένα μεγάλο εργοστάσιο θερμικής, ε, παραγωγής θερμικής ενέργειας που μολύνει ιδιαίτερα την περιοχή. Υπάρχει και μια μεγάλη εγκατάσταση εξεργασίας ύδατος. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η εταιρεία δεν έχει καταβάλει καμία προσπάθεια να βρει εναλλακτική τοποθεσία για την οικοδόμηση αυτής ε, της μονάδας. Η κατάσταση όμως δεν θα ήταν τόσο άσχημη αν η εταιρεία, ενώ παρουσίαζε το έργο στο Δήμο, είχε απαντήσει σε μία σειρά ερωτημάτων των πολιτών. Καταρχήν, τι γίνεται με τη διαλογή των αποβλήτων ε, και ε, ποιο ποσοστό των αποβλήτων θα αποτεφρωθεί. Δεν απάντησε επίση σε σχέση με τι τεχνολογίε που θα χρησιμοποιούνταν. Έτσι λοιπόν οι περισσότερε ερωτήσει ε, έμπαιναν αναπάντητε. Γι' αυτό το λόγο ήταν πάρα πολύ ταραγμένοι οι πολίτες, πιστεύω, πως όταν ε, κατασκευάζονται τέτοιες μονάδες ε, πρέπει οι πολίτες ε, να ενημερώνονται εκτεταμένως. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την δική μας επιτροπή που ανέλησε ταχεία την αίτησή μου, τη δική μου αναφορά. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Επίσης, θέλω να δράξω την ευκαιρία για να θέσω μια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με την Κομισιόν για περισσότερες πληροφορίες για το αν ήρθε και έρθει σε επαφή η Κομισιόν με τη Λιθουανική Κυβέρνηση για το ζήτημα αυτό ή όχι. Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα στην επικοινωνία μας με την Κομισιόν. Και μέχρι τώρα μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε μόνο με τη γραμματεία της ε, ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ Περιβάλλοντος. η εταιρεία και οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης πιστεύουν τώρα ότι θα πρέπει να απαντήσουν στην Κομισιόν. Έτσι λοιπόν, το τμήμα, το αρμόδιο τμήμα περιβάλλοντος του Δήμου έχει αναστείλει τη διαδικασία, γιατί κατάλαβε ότι ένα τέτοιο έργο δεν θα είναι δυνατό να τεθεί σε εφαρμογή χωρίς να έχει γίνει κάποια ανάλυση. Και τώρα θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν να μας δώσει μια γραπτή απάντηση σε σχέση με τις απαντήσεις ε, που έχει λάβει από τη Λιθουανική κυβέρνηση. Εμείς μέχρι τώρα δεν έχουμε λάβει τίποτα από την Κομισιόν. Φοβάμαι λοιπόν ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά, γιατί θέλουμε να δοθούν ε, καθολικές απαντήσεις ε, για τις σκοπούμενες δράσεις με αυτό το έργο, για να αποφύγουμε παρόμοιες περιπτώσεις στο μέλλον. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε σε εταιρείε να κερδίζουν εις βάρος της υγείας των πολιτών μας. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο από την Κομισιόν. Να σας πω ότι μας πιέζει ο χρόνος, γιατί θα πρέπει να συνεδριάσουν ε, οι συντονιστές. Παρακαλώ λοιπόν να είστε όλοι σύντομοι, γιατί δεν έχουμε, γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο που είχαμε για την Επιτροπή. Κύριε Βάιδα. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είμαι σύντομος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ε, Ευρωβουλευτή για την παρουσίασή του. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εξέτασε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω προσφυγής ε, που έθετε τις ίδιες ανησυχίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολούθησε πάρα πολύ, καλά, πάρα πολύ στενά τις περιβαλλοντικές, τα περιβαλλοντικές πτυχές. 19 του 2010 ενημερώθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είχε ξεκινήσει μια διαδικασία ε, Αξιολόγηση αντικτύπου ότι ολοκληρώθηκε και όπως αναφέρθηκε και από τον Ευρωβουλευτή στις 9 ε, Νοεμβρίου 2010 ε, ελήφθη απόφαση στη Λιθουανία ε, απόρριψης του περιφερειακού, της περιφερειακής εγκατάστασης αποτέφρωσης. Επομένως δεν δόθηκε τελικά η έγκριση, δεν δόθηκε η άδεια. Δεδομένου ότι εξακολουθεί να υφίσταται το θέμα της αναφοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι, δεν, ότι, ότι υπάρχει λόγος να συνεχίσει η έρευνα αν, ε, το, αν ο Ευρωβουλευτή έχει ε, περαιτέρω ε, ενημέρωση και στοιχεία για το θέμα. Ε, παρακαλούμε πολύ να έρθει σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Κύριος Παστινάρου, έχει ζητήσει το λόγο. Κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Μια Πρώτον, με εκπλήσει ότι ένα κράτος μέλος δείχνει μία τέτοια αδιαφάνεια προς τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές και δεν δίνει καν στον ε, ετώντα ε, τα αναγκαία στοιχεία για την αναφορά του που είναι μια στοιχειώδης υποχρέωση ενός κράτους μέλους. Προφανώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο για το θέμα της, ε, του Βίλνιους. Επίσης ε, χαίρομαι που δόθη μια τέτοια άδεια, αλλά ποιο είναι το συμπέρασμα από αυτή την κατάσταση. Διότι ε, θα επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή Προφανώς ε, οι, οι οδηγίες και οι νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ωραίες είναι, αλλά δεν είναι αποτελεσματικές. Θα έπρεπε λοιπόν να ενημερώσουμε ε, την, ε, τις αρχές της Λιθουανίας για την έλλειψη διαφάνειας και την ε, άρνηση ενημέρωσης του ενδιαφερομένου του θέματος. Ευχαριστώ. Ο αναφέρον έχει το λόγο. Σας παρακαλώ για δύο λεπτά σύντομα, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι στα όσα ακούσαμε από την Επιτροπή, από τον κύριο Μποστινάρο. Πρόεδρε. Χάρηκα πολύ που άκουσα την απάντηση από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν και ελπίζω να συνεχίσουμε τις συνεργασία μας στο μέλλον και ότι θα είναι και καρποφόρο. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Και εμείς το ελπίζουμε. Ευχαριστούμε και το συνάδελφο και αναφέροντα. Και αν κατάλαβα καλά, συνεχίζει να παραμένει ανοιχτή αυτή η αναφορά, αν κατάλαβα καλά. Λοιπόν, να κλείσουμε εδώ την ημερησία διάταξη και σε τρία λεπτά θα περάσουμε στη συνεδρίαση των συντονιστών. Σε τρία λεπτά θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών.